Κυρίε και κύριοι, ας ξεκινήσουμε ένα λεπτό μετά τις 3. Να σας καλωσορίσω, κυρίως να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας από το Βιετνάμ. Έχετε όλοι λάβει την ημερήσια διάταξη. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αιτήματα τροποποίησεων. Επομένως, γκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 2 έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων συνήθως. Το σχέδιο των πρακτικών των συνεδριάσεων της 6ης και 7ης Νοεμβρίου εγκρίνονται εκτός και αν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης. Σημείο 3. Οι αποφάσεις των συντονιστών στις 6 Νοεμβρίου και πάλι εγκρίνονται, εκτός και αν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι τα τέλη της συνεδριασής μας. Σημείο 4. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχουμε μία συνεδρίαση που αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο. Επομένως μπορούν όλοι να ακούσουν τα σχόλιά σας και τις θέσεις σας και να καλωσορίσω ίσως και όσους μας ακούνε στο Βιετνάμ και στη Λισαβόνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Τάλιν. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να μιλούν οι συνάδελφοι αργά για να μπορούμε να έχουμε και τη διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Σημείο 5. Πριν δύο χρόνια νομίζω υιοθετήσαμε ένα κανονισμό σχετικά με την κατανομή δεσμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ των 27 κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πριν ένα χρόνο, διορθώνει ο Πρόεδρος. Και υπήρξε ένα μικρό λάθος στο όλο εγχείρημα υπήρχε ένα σφάλμα σχετικά με την ποστόσωση ζάχαρης μεταξύ Ινδονησίας και Ινδίας. Έχουμε μία διαφορά ενός γράμματος στον κώδικα της χώρας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εντός ε, 24 ώρων αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, τότε θα εγκριθεί αυτή η τροποποίηση. Ως διορθωτικό στον κανονισμό. Θέλει κάποιο το λόγο? Όχι. Ευχαριστώ λοιπόν και την Γάμα Δελτάγκρη που είναι εδώ. Και φυσικά το κύριο θέμα σήμερα το απόγευμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με το εμπορικό επιμελητήριο στο Βιετνάμ για την ε, συμφωνία, την εμπορική συμφωνία και τη συμφωνία προστασίας και την ε, αλλαγή του εργατικού κώδικα. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο του Βιετνάμ. Ε, είναι εδώ ο πρόεδρος, κ. Σωτηράκης. Καλωσορίσατε. Και φυσικά θα έχετε και τη δυνατότητα να πάρετε το λόγο για τις ε, εμπορικές σχέσεις ε, και για τον ε, εργατικό κώδικα. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος εδώ, υπάρχει πολύ αριθμή την προσωπία. Καλώς ορίσατε. σας δώσουμε φυσικά το λόγο, αν το επιθυμείτε. Τώρα, για τον εργατικό κώδικα και των ε, τριών εκκρεμών συμβάσεων ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Ε, ο διευθυντής της ΔΟΕ, ο κύριος Αγκλή, είναι εδώ, του τμήματος της ΔΟΕ στο Βιετνάμ και φυσικά είναι και εμπειρογνώμονας ε, στις σχέσεις με το Βιετνάμ. Έχουμε και ε, μια αντιπροσωπεία, έναν ε, αντιπρόσωπο από την Συνομοσπονδία των Συνδικάτων και αυτός είναι εμπειρογνώμονας, είναι ειδικό για το Βιετνάμ και συμμετείχε και στη αντιπροσωπεία στο Βιετνάμ πριν από λίγες εβδομάδες. Να δώσω το λόγο λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Βιετνάμ. Ε, ο εισηγητής δεν είναι εδώ. Έχει αργήσει. Κύριε να έχει καθυστερήσει η πτήση του. Θα έρθει, θα έρθει, αλλά ζητά συγγνώμη γιατί έχει καθυστερήσει η πτήση. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, για 12 λεπτά, ο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Μιλητηρίου. Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είμαι πολύ ευτυχής. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ. Είναι η πέμπτη φορά που παίρνω το λόγο την τελευταία φορά μίλησα πριν από λίγε εβδομάδε στο ΑΝΟ. Είμαι πολύ ευτυχή σήμερα που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ο Νικολά Οντιέ. Είμαι δικηγόρο, νομικό και από το 1993 συμμετέχω στι ε, δραστηριότητε του εμπορικού επιμελητή, ιδιαίτερα σε αυτέ που έχουν σχέση με την Ασία και το Βιετνάμ. Από το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων ε, ήμουν παρών. Θα ήθελα να σας πω το Ευρωπαϊκό εμπορικό επιμελητήριο, το Eurocham και επειδή ήρθαμε με μεγάλη, αν θέλετε, αντιπροσωπεία, εκπροσωπείται το Βιετνάμ, χίλια μέλη συγκεκριμένα εκπροσωπούνται, χίλιες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες, καθώς και μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε να βελτιώσουμε το περιβάλλον των εμπορικών σχέσεων, των επενδύσεων, για ο κάθε είδους επιχειρήση στο Βιετνάμ έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια και παρακολουθούμε τις πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει από το 98 και πέρα το 97 όταν άνοιξαν για πρώτη φορά οι πόρτες ε, του εμπορίου από την κυβέρνηση στο Βιετνάμ. Αναφέρομαι εδώ σε πολύ σημαντικές ε, ε, μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε πολλές περιοχές και αυτό σε όλες τις περιοχές ε, του Βιετνάμ και θα ήθελα εδώ να συμπεριλάβω σε αυτό όλα μας τα μέλη. Έχουμε από όλους τους τομείς, από την αυτοκινοβιομηχανία, τα ενοπνευματόδη, την ε, βιομηχανία σε όλους τους τομείς υψηλού επίπεδου τεχνολογία και έχουμε επαφές με τα Υπουργεία στο Βιετνάμ Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου και βεβαίως τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε επαφές όχι μόνο με αξιωματούχους της κυβέρνησης των περιφερειακών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των διευθυντών των μεγάλων επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε φυλάδια και έγγραφα τα οποία αναφέρονται ουσιαστικά στην θέση και την τοποθέτηση των χιλίων μελών μας. Τις τελευταίες δεκαετίες, από τότε που ξεκίνησε το πρώτο κύμα των ε, επενδύσεων στο Βιετνάμ, ο τομέας είναι ζωντανός και μεταρρυθμίζεται διαρκώς. Από το 1992-1993 μέχρι σήμερα πρόκειται για μια διαφορετική χώρα. Όλα έχουν αλλάξει. Και αυτό, ακριβώς επειδή υπάρχουν επενδύσεις, επειδή υπάρχει παρουσία των ευρωπαϊκών επενδύσεων και των ευρωπαϊκών αξιών. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του μεγάλου προγράμματος ε, των ε, επενδύσεων αλλά και των συγκεκριμένων προγραμμάτων επενδύσεων μέσω των δωρητών βοηθήσαμε τη χώρα αυτή να εξελιχθεί, να μεταρρυθμιστεί, καταρχήν μέσω μεγάλων επενδύσεων στις υποδομές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και βεβαίως ε, μέσω του νέου κύματος επενδύσεων που έχει επιταχύνει ακόμα περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε ένα νέο ε, κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ της ε, Ευρώπης και του Βιετνάμ. Έχουν υπογραφεί πάνω από 60 εμπορικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και η Ευρωπαϊκή επενδυτική δραστηριότητα η οποία έχει ενισχύσει όχι μόνο τις υποδομές αλλά όλους τους τομείς ε, των ελεύθερων συναλλαγών. Εμείς ε, μέσω της δικής μας ε, οργάνωσης στηρίζουμε τις επενδύσεις αλλά όχι μόνο και την εξέλιξη των κοινωνικών δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσω αυτών των συμφωνιών και με νέε συμφωνίε οι οποίες επεξεργαζόμαστε και θα υπογραφούν διαπιστώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην αφήσουμε αυτήν την αγορά να καθυστερήσει. Ξέρετε ότι η μεγάλη ανταγωνιστή είναι η Κίνα, η Κορέα και η Ιαπωνία. Σήμερα το Βιετνάμ βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Η Το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο σήμερα θα χρησιμοποιήσει μέσω της Συμφωνίας ε, Ελεύθερων Συναλλαγών της ε, μέχρι σήμερα διμερείς ε, συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί νομικοί εργάζονται και οι περισσότεροι που θέλουν σήμερα να επενδύσουν, οι περισσότεροι πελάτες μας, όλοι αυτοί που περνάνε μέσα από το εμπορικό επιμελητήριο, θέλουν να ξέρουν ποιες είναι οι προστασίες και ποιες είναι ε, οι ε, δυνατότητες προστασίας που έχει ένας επενδυτής. Ανοίγουμε λοιπόν νέα κεφάλαια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται, που είναι ήδη παρόντες στο Βιετνάμ, ε, πρόκειται για την ορθή υλοποίηση αυτής της συμφωνίας διμερής διάλογος και η παρουσία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ε, ομαλή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρώπης και του Βιετνάμ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα συμβούλιο που θα βρίσκεται στην καρδιά αυτών των επενδύσεων, ένα συμβούλιο μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκών Ενώσεων, έτσι ώστε να υπάρξει υπεραιτέρω ομαλή υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Βεβαίως θα πάρει χρόνια και ξέρουμε σήμερα ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργήσει σωστά στην πράξη αυτή η συμφωνία. Όπως σας είπα από την αρχή, αυτή η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα βοηθήσει τους ε, ε, συμμετέχοντες να καλύψουν τα κενά. Θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, αλλά και τους ε, ηγέτες, τους συμμετέχοντες από την πλευρά του Βιετνάμ, οι οποίοι περισσότεροι έχουν περάσει από πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στην Αμερική, να υλοποιήσουν με έναν θετικό τρόπο αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία θα κάνει κάτι παραπάνω από το ενισχύσει και να επιταχύνει τις ε, υπάρχουσες επενδύσεις. Θα βοηθήσει έτσι ώστε να ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, να ενισχυθεί ο εργατικός κώδικας και βεβαίως να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσω της συμφωνίας αυτής για να ενισχύσουμε την προστασία τους. Βλέπετε ότι η Κίνα ενδυναμώνει την ε, θέση της. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν κάνει κάτι παραπάνω, η Κίνα θα παίξει ακόμα πιο ε, καθοριστικό ρόλο στην περιοχή. Τα μέλη μας γνωρίζουν ότι η δική μας τοποθέτηση είναι καθοριστική. Θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Το 2019 ξεκινήσαμε μια, ένα σύστημα παρακολούθησης ε, των μελών μας. Πάνω από το 80% απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών βοηθάει την βελτίωση όχι μόνο των οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανοίξουμε το νέο κεφάλαιο των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ και πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους στόχους. Θα δώσω αμέσως το λόγο στους συναδέλφους γιατί υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά μηνύματα τα οποία πρέπει να διοχετεύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συναδελφοί. Ονομάζομαι Χάν και είμαι η μέρα του Eurojump. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα κάποιε πρόσφατε εξελίξει ό,τι αφορά το εργασιακό δίκαιο στο Βιετνάμ. Ξέρουμε λοιπόν ότι η εργασία και η απασχόληση αποτελούν βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη Σύμφωνη Ελευθέρω Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένη και τη EVFTA. Θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι θέλουμε να τονίσουμε την δέσμευση του Βιετνάμ σε ό,τι αφορά τη συμφωνία και το Βιετνάμ λοιπόν στι 20 ε, Νοεμβρίου του 2019 πέρασε μια καινούργια νομοθεσία και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2029. Και έχουμε και άλλες εξελίξεις ότι αφορά την ε, επικύρωση της σύμβασης ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Θεωρούμε λοιπόν τον νέο κώδικα του 2019 μια μεγάλη πρόοδο και Θεωρούμε ότι αυτό αντιπροσωπεύει τις προσπάθειες του Βιετνάμ να εντοπίσει και να εντάξει τις εργασιακές συνθήκες υπό την ΠΟΕ ε, στο εργασιακό του δίκαιο. Το Βιετνάμ είναι μια περιοχή που έχει περάσει πολλές αλλαγές λοιπόν υπέρ του εργοδότη με μεγάλες αλλαγές και νέα νομοθεσία που προστατεύει περαιτέρω τα δικαιώματα των εργαζομένων και προσαρμόζονται στα διεθνή πρότυπα. Και δεν θα περάσω λοιπόν σε επίπεδο μεγάλε λεπτομέρειε ό,τι αφορά τι αλλαγέ, αλλά να τονίσω κάποια βασικά ζητήματα υπό τον κώδικα. Καταρχά, ε, ο οριακό κώδικα εισαγαγεί νέε ρυθμίσει που προσαρμόζουν ε, τα πρότυπα σε ό,τι αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσαι και την προστασία των ε, εργαζομένων να οργανώνονται και να συνδικαλίζονται σύμφωνα με την συνθήκη του ΠΟΕ. Επίσης, το δικαίωμα των εργαζομένων πέρα από την ε, συνδικαλίζεστε να δημιουργήσουν, να καθορίζουν εκπροσώπους και αντιπροσώπους των εργαζομένων σε τέτοια συμβούλια. Και σύμφωνα με το νέο αυτό σύστημα, τα ανεξάρτητα συνδικάτα θα έχουν τέτοια δικαιώματα και υποχρεώσεις και ακριβώς τις ίδιες ευθύνες. Προ του εργαζόμενου και του εργοδοτέ. Κατά δεύτερον, ο κώδικα του 2019 εισήγαγε ρυθμίσει για να διευκολύνει την επίλυση εργασιακών διαφωνιών ε, με την ε, συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών. Επίσης, ε, ρυθμίσεις για την καταγκαναστική εργασία σε ό,τι αφορά τον σαφή ορισμό του εξαναγκασμού σε εργασία και επιτρέπουν στους εργαζόμενους μονομερά, μονομερός να καταργήσουν και να την άμα, ε, και σύμβαση χωρίς να τη δικαιολογήσουν και επίσης ε, οι επιθεωρητές εργασίες μπορούν να κάνουν αυτήν επιθεωρήσεις για να ελέγχουν θέματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τη ζωή, την υγεία, την ε, τιμή και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στον χώρο εργασία. Επίση, ε, περιλαμβάνονται πολλέ ρυθμίσει για την παιδική εργασία, σε ό,τι αφορά επίση ε, την απασχόληση. Έχει επικυρωθεί πλέον η σύμβαση του που υπαριθμών 100 και 111 για την διακριτική μεταχείριση. Επίσης, το δίκαιο του Βιετνάμ πλέον είναι πολύ εκτενές σε ό,τι αφορά την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Επίσης, ε, τονίζουμε την ίση ε, μεταχείριση των γυναικών. Και δεν υπάρχει δυνατότητα απλά να υπάρχει κατάλογος ε, ε, απασχόλησης για, που απογορεύεται τις γυναίκες. Επίσης, ε, θα θέλαμε να σας πούμε ότι στις 15 Ιουνίου του 2019 το Βιετνάμ επικύρωσε τη Σύμβαση 198 για τις συλλογικές συμβάσεις, την υπερθμό 98. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι πλέον υπάρχει επικύρωση 6 συμβάσεων στο δίκαιο του Βιετνάμ και από πλευρά μα το Βιετνάμ δεν κάνει λιγότερα από τη Σιγκαπούρη και το, άμα, η Ιαπωνία οι δύο χώρες αυτές ε, επικύρωσαν επίσης έξι βασικές συμβάσεις ε, του ΠΟΕ. Βρισκόμαστε λοιπόν στο ίδιο επίπεδο. Ο πήγης είναι στο ίδιο επίπεδο όπως και οι άλλες δύο χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λέγει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για την επισκόπηση αυτή. Και τώρα να ακούσουμε και την πλευρά του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό του εργασιακού κώδικα. Ο κύριος Λί και ο κύριος Μάιερ. Για 12 λεπτά Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας που καλέσατε το ΔΟΕ σε αυτή τη σημαντική συνεδρίαση. Ε, εδώ εκπροσωπείται από τον κύριο Ντεμάιερ που έχει εργασιστεί τα τελευταίους δύο γύρους της μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου το 12 και το 19 και είναι τώρα ανώτερος ε, σύμβουλος ε, ε, στο Διεθνές Τμήμα ε, Προτύπων Εργασίας. Εγώ λέγομαι Τσανκλή, εργάζομαι στο Ανόη από το 2015. Ε, είμαι διευθυντής στη ΔΟ και έχω εργαστεί σε βιομηχανικές σχέσεις και στο εργατικό δίκαιο τα τελευταία 19 χρόνια φέτος με την κύρωση της σήμερα 98 του Ιούνιου και την υιοθέτηση του νέου εργατικού κώδικα στις 20 Νοεμβρίου που θα ε, εισαγάγει αρχές του δικαιώματος του συνεστερίζεστε σε επίπεδο επιχειρήσεων και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο βιομηχανικών σχέσεων στο ουσιαστικό Βιετνάμ. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητούμε την απόφαση του Πρωθυπουργού για το σχέδιο δράση ε, να ε, επικυρώσει τη συμβάση 105-2020 και την 87 το 2023 στο πλαίσιο της ε, παγκόσμιας ολοκλήρωσης ένταξης του Βιετνάμ μέσω της ε, Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών, κυρίως ε, μέσω της Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και της CPTTP. Μέχρι το 2014 δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το Βιετνάμ θα πάει τόσο μακριά όταν ξεκίνησα το έργο μου στις αρχές του 2000, κανένα στο Βιετνάμ δεν καταλάβανε τι σήμαιναν οι βιομηχανικές σχέσεις, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση. Έπρεπε να ξεκινήσουμε την βασική κατάρτιση για να βοηθήσουμε ε, τον κόσμο να καταλάβει τις βασικές έννοιες και να απτύξουμε ορολογία στα βιετναμέζικα. Μόνο τότε αρχίσαμε να διευρύνουμε νέους τρόπους ε, διαχείρισης των κοινωνικών σχέσεων. Όμως ο όρος ελευθερία του συνεταιρίζεστε, δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, έμενε ταμπού μέχρι το 2014 και θεωρείται συνώνυμο με την πολιτική ανατροπή ήταν ε, πραγματικά η TTP σήμερα, η Συνολική και Προθετική Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού και τώρα η ε, Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που άνοιξε ε, την ε, συζήτηση για το δικαίωμα τη συνειστερής και άλλε αρχέ δυνάμει τη δήλωση ΕΔΟΕ για τι θεμελιώδει αρχέ και τα δικαιώματα στην εργασία. Όταν αποσύρθηκαν οι ΗΠΑ από την TTP το 2017, οι περισσότεροι στο ΕΝΟΗ πίστεψαν ότι είχε πεθάνει το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων ε, μαζί ε, με τα κίνητρα για την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ. Όμω, αναζωογονήθηκε το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων και είδαμε πρόοδο το 2019. Πρέπει να πω ότι η επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας υπό τον κύριο Λάγκη το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν πολύ σημαντική στο να ζωγονήσει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Και σε εσωτερικό επίπεδο, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έδωσε φωνή στου ισότητε των μεταρρυθμίσεων που πάντοτε αναγνώρισαν ε, ότι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι και το δικαίωμα στι συλλογικέ διαπραγματεύσει ε, ε, πρέπει να υπάρχει στο, στο Βιετνάμ από τις αρχές του 2000. Όμως ε, υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί και στην κυβέρνηση και στο κόμμα, στην Εθνοσυνέλευση, στα συνδικάτα. Η συμφωνία τους βοηθά να αποκτήσουν επιρροή εντός του συστήματος και να σημειώσουν τις πρόοδους που είδαμε φέτος. Επίσης, πρέπει να αναφέρω τον κριτικό ρόλο που έπαιξε συνδυασμό στενού συντονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τη ΔΟΕ και των Βετναμέζων εταίρων ε, στο να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση στο ψηλότερο επίπεδο ε, πολιτική λήψη αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα παρήχαν πολιτική στήριξη σε καθημερινή βάση. Ε, η σύμπραξη που βασίζεται στο σεβασμό στην εμπιστοσύνη και στην υπομονή και ο αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ΔΟΕ και Βιετναμιζική Κυβέρνηση είναι που, αυτό που έκανε τη διαφορά στο να προωθηθούν ε, τα εργασιακά δικαιώματα δυνάμει τη συμφωνία. Οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη δεν έχουν παράξει το επίπεδο πρόοδου, αυτής πρόοδου για να κινηθούμε προς ε, την κύρωση της ε, σύμβασης της ΔΟΗ υπερθμών 8. Ε, φυσικά, έχουμε για την Κορέα 4, για την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη 6 ακόμη. Φυσικά, το Βιετνάμ ε, πιστεύω ότι του χρόνου θα επικυρώσει και την Σύμβαση 87 και ελπίζουμε μέχρι το 2023 να επικυρώσει και τη Σύμβαση 87. Θέλω να ευχαριστήσω όμως την υποστήριξη της ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ εμπορίου γιατί πραγματικά ε, υποστήριξε τους κοινωνικούς εταίρους στο Βιετνάμ. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις ενωπιών μας, ε, κυρίως ε, η Σύμβαση 87 για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε, η οποία θέτει ένα ενδιαφέρον θέμα συμβατότητας μεταξύ του δικαίωματος του συνεταιρίζεσθε για των ειδικών αρχών και του σοσιαλιστικού πολιτικού συστήματος. Όμως είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο θα κυρώσει τη σύμβαση του Βιετνάμ, αλλά θα προχωρήσει και στην εφαρμογή της. Αν δείτε το κείμενο του υιοθετημένου εργατικού κώδικα, έχουμε βελτιώσει στις διατάξεις για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση 98 και εισάγονται και αρχές του δικαιώματος της συνεταιρίζεσης στις επιχειρήσεις. Ε, σε μικρό βαθμό, αλλά αρκετά σημαντικό. Αυτή η αλλαγή αποτελεί πολύ μεγάλη πρόοδο που μπόρεσε να κάνει η χώρα το 2019 βάσει πολιτικού συμβασμού που έγινε στο πολιτικό γραφείο ε, που είναι το ανώτατο πολιτικό σώμα στο Βιετνάμ. Όμως ε, το Βιετνάμ, αυτές οι αλλαγές που έγιναν το 2019 αρχίζει να ακολουθεί ένα πραγματικά διαφορετικό δρόμο από την Κίνα στο θέμα της ε, ανάπτυξης. Ναι, βέβαια έχουν αφαιθεί και κάποια θέματα για μελλοντικές ε, συζητήσεις. Ε, το 2021 όμως πιστεύω ότι θα έχουμε ανεξάρτητες οργανώσεις εργαζομένων που θα αρχίσουν να συνδέονται ή να συνεταιρίζονται με άλλους. Και ε, θα τους ε, παρέχουμε στήριξη το 2021 πέρα από το επίπεδο της επιχείρησης. Και πρέπει να πω ότι δεν θα είναι εύκολο για το Βιετνάμ ε, να επαναχωρήσει την πρόοδο όταν θα έχει προχωρήσει για τους εξή λόγους. Μέχρι το 2018 το Βιετνάμ είχε λίγες διεθνείς υποχρεώσεις, όμως η κατάσταση θα διαφέρει από το 2021 και μετά. Καταρχήν η TPP ισχύει από τον Ιανουάριο του 2019. Δεσμεύεται λοιπόν από τη σύμβαση αυτή του Βιετνάμ. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την κύρωση της ε, Σύμβασης 98, οι εποπτικέ αρχές της ε, ΔΟΕ πιθανότατα ε, θα κάνουν τα πρώτα του σχόλια για την εφαρμογή. Ε, τουλάχιστον να έχουμε την πρώτη έκθεση από την κυβέρνηση του Βιετνάμ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021. Ε, τρίτον, αν επικυρωθεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε μια σειρά ε, διαλόγου εποπτείας ε, και φορέων διευθέτησης διαφορών. Πιστεύω ότι αυτά τα πολλαπλά στρώματα εποπτείας θα κρατήσουν το Βιετνάμ στην πορεία του προς το να σεβαστεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Εδώ έχει δύο εντολές, έχει διπλή εντολή Καταρχήν, ε, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να γίνουν σεβαστέ σύμβαση 98 και 87. Δεύτερον, θα παρέχει υποστήριξη στου εθνικού εταίρου, ε, προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση για το νέο σύστημα που θα βασίζεται στι λογικέ διαπραγματεύσει και στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Και πιστεύω ότι με τη δική σα υποστήριξη και τον ενεργό ρόλο που να παρέχετε βοήθεια και να παρέχετε και εποπτεία, θα βοηθήσετε ιδιαίτερα τη ΔΟΕ να υιοθετήσει το θεματολόγιο αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Ναι, πιστεύω ότι ο θετικός αντίκτυπος ε, της ε, Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ ε, Παρέχει πολιτική δέσμευση ε, για τα διεθνή εργατικά τρόποτυπα και είναι κάτι απτό. Ε, ακόμη και πριν την επικύρωση της ε, συμφωνίας έγιναν διάφορες αναφορές ε, το 2000, στη σύμβαση του 1998, όμως το 2019 το Βιετνάμ κύρωσε τρεις συμβάσεις εδώ σε σχέση με την αποκατάσταση των ανθρώπων με αναπηρίες σε σχέση με τις υπηρεσίες ε, δημόσιες, ε, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και πιο πρόσφατα την 98 που ε, έχει να κάνει με την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτές οι κυρώσεις ήταν η από το 2014 και συμπεριλάμβανε την πρώτη επικύρωση μια θεμελιώδης σύμβαση από τότε που επικυρώθηκε το 2007 η Σύμβαση για την Κατεδανικαστική Εργασία φτάνουμε στον αριθμό 24 ε, για το Βιετνάμ ε, σε ό,τι αφορά την επικύρωση ε, διεθνών συμβάσεων βρίσκεται ουσιαστικά στο μέσο όρο για την περιοχή Ασίας Ειρηνικού που διστάζει ουσιαστικά να επικυρώσει τέτοιε συμφωνίε. εδώ το Υπουργείο Εργασία του Βιετνάμ συνεργάζονται σε μια στρατηγική 30 ε, ε, με 30 που πιθανότατα θα σημαίνει ότι μέχρι το 2030 το Βιετνάμ θα επικυρώσει 30 συμβάσεις και 8 ε, συμβάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μεταξύ αυτών έχουμε και τεχνικά πρότυπα που σχετίζονται με τον ελάχιστο μισθό, ελάχιστα πρότυπα για την κοινωνική ασφάλιση και την αξιοπρέπεια εργασία για τους αλείς. Και καθώς τώρα αυτά είναι από εξέταση, το γενικό, οι συμβάσεις γενικού πλαισίου της ΔΟΕ για την ασφάλεια και την ε, υγεία στην εργασία, δηλαδή 155-117 θα πρέπει να γίνουν θεμελιώδεις συμβάσεις και ήδη αυτές τις έχει επικυρώσει το Βιετνάμ. Είναι σαφές ότι με την επικύρωση και την εφαρμογή φυσικά της Σύμβασης 87 και της 105, παραμένουν δύο δηλαδή, τον επόμενο των δύο που παραμένουν μπαίνουμε πολιτικά σε μια φάση μεταρρυθμίσεων με ιδιαίτερες ε, προκλήσεις, ε, γιατί αυτά αφορούν κυρίως ε, τις πολιτικές ελευθερίες και τα πολιτικά δικαιώματα. Και αυτές οι ελευθερίες και τα δικαιώματα συνεχίζουν να προκαλούν αμφιβολίες για την πολιτική βούληση για μεταρρύθμιση. Ο εργατικός κώδικας που υφετήθηκε πρόσφατα ανοίγει την αρένα των εργασιακών σχέσεων σε ε, εκπροσώπους από τα κάτω, όπως αποκαλούνται, σε επίπεδο επιχείρησης. Αλλά φυσικά η μεταρρύθμιση δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι να υπάρξει αναθεώρηση του νόμου περί συνδικάτων και της σύστασης ε, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας του Βιετνάμ, ε, η οποία κρατά τα προνόμια που έχει κερδίσει ως μέρος του κινήματος που οδήγησε στην απελευθέρωση και στην εθνική κυριαρχία του Βιετνάμ. Τι θα κάνει τώρα εδώ, ε? θα συνεχίσει να προωθεί την επικύρωση της Σύμβασης 87 και αν είναι δυνατό πριν από το 2021. Αυτό προκειμένου να διασφαλίσουμε την ε, πρόοδο που βλέπουμε ότι γίνεται με την ε, υιοθέτηση του εργατικού κώδικα. Εδώ επίσης θα βοηθήσει στην κατάρτιση των εκτελεστικών κανονισμών ε, του εργασιακού κώδικα. Πολλές λεπτομέρειες θα πρέπει τώρα να καταρτιστούν περαιτέρω. Και επίσης θα ασχοληθούμε με την λεπτομερή καταγραφή δικαιωμάτων ε, σε ό,τι αφορά την συλλογική εκπροσώπηση. Επίσης, ε, εδώ θα παρακολουθήσει έναν αυξανόμενο αριθμό ανεξάρτητων εκπροσώπων ε, οργανώσεων, εκπροσώπων εργαζομένων και επιθυμούμε να εγγραφούν στο Υπουργείο οι οργανώσεις αυτές. Επίσης, θα παρακολουθούμε αν ε, οι ανεξάρτητες αυτές οργανώσεις μπορούν να ανταγωνιστούν για δικαιώματα συλλογικών διαπραγματεύσεων με, τις, με τα συνδικάτα που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων και αν ε, επιτροπές ε, δεν έξιων θα μπορούν να επιλύουν τέτοιες διαφορές. Και εδώ θα ευχαριστήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και ο συνάδελφος για την υποστήριξη που έχει δώσει στη ΔΟΕ και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να μας παρέχεται αυτή την υποστήριξη. Η κύρωση της Σύμβασης 105, άλλη θεμελιώδη σύμβαση που έχει να κάνει με την καταναγκαστική εργασία, είναι πολύ σημαντική καθώς θα απαγορεύσει στο Βιετνάμ να χρησιμοποιείται καταναγκαστική εργασία ε, έναν μέσο πολιτικού καταναγκασμού ή εκπαίδευση ή τιμωρία για την έκφραση πολιτικών απόψεων ε, ή απόψεων ε, που ε, είναι αντίθετες με το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό κατεστημένο. Και η κύρωση θα αποτελέσει ένα τεστ για την εξέλιξη προς μεγαλύτερες πολιτικές ελευθερίες, πιστεύουμε ότι το Βιετνάμ θα επικυρώσει του χρόνου αυτή τη σύμβαση ήδη το 2007 είχε τεθεί η προσωπική ρωσή σύμβαση, αλλά την ε, τελευταία στιγμή αποσύρθη. Και μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό σχετιζόταν με φόβους ε, για καταδίκη σε σχέση με το σεβασμό πολιτικών ε, δικαιωμάτων. Ο τοπικό κώδικα του Βιετνάμ τροποποιήθηκε το 2015 και ε, κατέστησε ποινικά κολάσιμο αδίκημα την καταναγκαστική εργασία, επιβάλλοντα πρόστιμα από 2.800 ευρώ και ποινικά κάθεξη από 6 μήνε ω 12 χρόνια. Και αυτό θεωρήθηκε πρόοδο δυνάμει τη Σύμβαση 29. Πιστεύουμε ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Βιετνάμ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Και αυτό σε διαφοροποίηση με παρόμοιες δεσμεύσεις Δυνάμει της CPTTP, η Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην επικύρωση των διεθνών εργασιακών προτύπων, δηλαδή ε, δεν μιλάμε μόνο για την υλοποίηση των θεμελιωδών ερχών, αλλά και της επικύρωσης των συμβάσεων. Επίσης, ε, δίνει σημασία στις τεχνικές ε, συμβάσεις ε, και καθιστά τη ΔΟΕ αντικειμενικά υπεύθυνη να παρακολουθεί τη συμμόρφωση. Καλωσορίζουμε την προσέγγιση αυτή. Ίσως βέβαια πρέπει να κινηθούμε προσεκτικά, γιατί οι εταίροι στο παρελθόν ήταν κάπως διστακτικοί και μιλάω γενικά για τέτοιους ε, συνεργάτες ήταν λοιπόν διστακτικοί να εφαρμόσουν ε, τις ε, ρήτρε περιεργασία στις συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσει τη μοχλευσή της πιο ενεργά από ό,τι στο παρελθόν αν επικυρωθεί η συμφωνία. Η πιο πρόσφατη θεώρηση του εργατικού κώδικα είναι το δεύτερο τμήμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια αφού μπήκε στον ΠΟΕ του Βιετνάμ Έχουμε δώσει εκτεταμένα σχόλια σε ένα προσωρινό σχέδιο και τα παρουσιάσαμε αυτά στην Εθνοσυνέλευση. Η συζήτηση μας δείχνει ότι υπάρχει βούληση να καλυφθούν τα κενά σύμφωνα με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όμως ε, υπάρχει και απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Πιστεύουμε ότι πέρα από το θέμα των συλλογικών δράσεων θα έχουμε αυτή τη διαδικασία περισσότερους εργαζομένους στην επίσημη οικονομία, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και το Βιετνάμ θα είναι πιο ισχυρό για να αντιμετωπίσει τη γυράση του πληθυσμού. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι συμφωνήσαμε για ένα χρόνο ομιλίας με κάποιες περιορισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παρόλα αυτά για όλες αυτές τις πληροφορίες και θα δώσω τώρα το λόγο στην Ομοσπονδία των ε, Συνδικάτων. Έχετε 7 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης ε, του Βιετνάμ καθώς ε, και τη βιωσιμότητα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Βιετνάμ, κάτι που έχει κυρωθεί πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει και για την 105 αλλά και για την 87 συμφωνίας η υπόσχεση για την κύρωσή της. Και βεβαίως η Συμφωνία 98 για τις συλλογικέ συμβάσεις, η οποία κυρώθηκε και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2018. Βάσει αυτής της συμφωνίας, ε, της Συμβασίας 98, οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί θα πρέπει πλέον να υλοποιηθούν και στην πράξη. Βάσει της ε, συμφωνίας C105 και C80 θα πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν ανακοινωθεί και επισήμως στην ε, Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Επιπλέον, πέραν δηλαδή αυτών των συμβάσεων, Υπάρχει η δέσμευση για την τήρηση της αρχής ε, των ε, συλλογικών συμβάσεων, της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Στην πράξη όμως δεν υπάρχει μια πραγματική πρόοδος και όσον αφορά την αρχή του συνεταιρίζεσαι, αλλά και όσον αφορά την, ε, ελευθερία που συνεταιρίζεστε και της ε, ελευθερίας ε, έκφρασης ε, αλλά και διαπραγματεύσεων, συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας πλήρης και αυστηρός έλεγχος των δικαιωμάτων αυτών, της προστασίας του σεβασμού της από μέρου των εθνικών αρχών και της κυβέρνησης. Και θα πρέπει βεβαίως να υπάρξει τήρηση αυτών των δεσμεύσεων σοβαρή παρακολούθηση και από μέρους των κοινωνικών εταίρων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεται και των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται και να γίνεται σεβαστό έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχουν φορείς αυτόνομοι για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, να τηρούνται οι δεσμεύσεις, ιδιαίτερα όλα αυτά που προβλέπεται στην ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Όλα αυτή η έλεγχη και επιτήρηση θα πρέπει να γίνονται και στο χώρο εργασίας, αλλά και γενικότερα στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για την τήρηση σωστών και βιώσιμων εργατικών και εργασιακών σχέσεων η αναγνώριση του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ένα θεμελιώδες δικαίωμα που θα πρέπει να τηρείται και το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θα πρέπει δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να επιλέξει να εκπροσωπείται από έναν συλλογικό φορέα, από μία συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία αναλαμβάνει την ε, συλλογική διαπραγμάτευση και αυτό βεβαίως δημιουργεί και ένα ε, φιλικό και επικοδομητικό κλίμα στις ε, εργασιακές σχέσεις. Βεβαίως, δεν υπάρχει εδώ καμία σαφής πρόβλεψη στα νομοθετικά κείμενα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο νόμος δηλαδή στο Βιετνάμ δεν προϋποθέτει την ίση εκπροσώπηση των εργαζομένων μέσω αυτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν είναι λοιπόν σαφής η σχέση στην ε, νομοθεσία, ούτε και οι διατάξεις που προβλέπουν ε, την ε, εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων την διεκπαιρέωση και τις διαδικασίες για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Χωρίς να υπάρξει προστασία των δικαιωμάτων της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι λειτουργεί η αγορά εργασίας και εργασιακές σχέσεις σεβόμενη την τήρηση των δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, η ασφάλεια, είναι κάτι που υπονομεύεται στην πράξη. Υπάρχουν δηλαδή νομοθετικά κενά. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Βιετνάμ, πάνω από 80 διατάγματα καλύπτουν αυτά τα κενά της εργατικής νομοθεσίας. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι συνεχίζει να μην λειτουργεί το σύστημα της εκπροσώπησης των εργαζομένων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με έναν απρόσκοπο τρόπο. Ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις, η λειτουργία τους, η δυνατότητά τους να προστατεύσουν τα κοινωνικά και δευτεριακά δικαιώματα των εργαζομένων, η τήρηση του δικαιώματος του συνεταιρίσματος, η ελεύθερη έκφραση, η ελεύθερη ε, δυνατότητα διαμαρτυρίας είναι δικαιώματα τα οποία δεν διασφαλίζονται. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να αποτελέσουν τμήματα των νέων μεταρρυθμίσεων, κάτι το οποίο περιμένουμε. Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης του συνεταιρίζεται, παρουσιάζουν αδυναμίες. Υπό αυτές τις συνθήκες η κατάσταση παρουσιάζεται ως επικίνδυνη. με τις ε, συνεχείς ε, μεταρρυθμίσεις σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι δύο συμφωνίες που εκκρεμούν και δεν έχουν ακόμα ε, κυρωθεί, η 7 και η CET8, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να επικυρωθούν. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν, ιδιαίτερα όσον αφορά την δυνατότητα καταγραφής των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων, της ε, επιθεώρησης και ελέγχου στον χώρο εργασίας, επίσης όσον αφορά την επίλυση διαφορών σε θέματα εργασιακών σχέσεων, μηχανισμούς για την σωστή ενημέρωση και τον έλεγχο όσον αφορά τις ε, εργασιακές σχέσεις. Επαναλαμβάνω, η CET7 και η C105, οι δύο αυτές συμφωνίες θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να κυρωθούν. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τεχνική βοήθεια και κάθε σύμβουλη σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και στις εθνικές αρχές και στην κυβέρνηση του Βιετνάμου. Ολοκληρώνω. Έχουμε δεσμευθεί έτσι ώστε να συνεχίσουμε την στήριξη των μεταρρυθμίσεων με σκοπό να προστατεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα και τα εργασιακό δικαιώματα των εργαζομένων στο Βιετνάμ. Σας ευχαριστώ και τώρα να ακούσουμε ε, και τη συζήτηση ο κύριος Μπουζουά, ο οποίος ε, ε, Αντικαθέτω τον ε, συγητή μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και αν με επιτρέψετε θα διαβάσω αυτά που μας έχει πει ο μόνιμος συγητής αξιότιμη Πρόεδρε Κυρίε και κύριοι και αγαπητοί προσκαλεσμένοι, χαίρομαι που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψε. ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή, όπου το τελικό σχέδιο και η επικυρωμένη μορφή των συμφωνιών ε, επέρχεται για το Βιετνάμ. Έχουμε τη ε, συνομιλήσει με κάποιους από εσάς ε, στην επίσκεψή μας στο Βιετνάμ την προηγούμενο μήνα, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και πιο πολλά. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τις πολύτιμες συμβουλές σας ε, και για την δουλειά που γίνεται, που θα πρέπει να γίνει και σωστά. Είναι πολύ σημαντικά να υπάρχει σωστή επικέντρωση σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο Βιετνάμ, σε ό,τι αφορά την ανάλυση του νέου εργασιακού κώδικα. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα νομικά και πρακτικά μέτρα ε, επιτόπου στο Βιετνάμ, τα όσα απαιτούνται και αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει το Βιετνάμ. Τρει ερωτήσει, λοιπόν έχει ο συνάδελφος κύριε Πρόεδρε. Καταρχά ε, προ την EU Chamber συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο. Οι επιχειρήσεις, μάλλον σε ό,τι αφορά την προσωρινή ε, εφαρμογή των συνθήκων. Ξέρουμε ότι πολλά έχουν γίνει, αλλά θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε σε ό,τι αφορά τις ε, συνθήκε, τι προκλήσεις και τις Ευκαιρίε που ενέχει αυτή η συμφωνία. Κατά δεύτερον, πόσο έχουμε προχωρήσει στην προετοιμασία στη σύσταση των ε, χώριων ε, συμβουλευτικών σωμάτων και σε ποια φάση βρίσκεται ο ΠΟΕ σε ό,τι αφορά τη δικασία αυτή προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνουμε κάποια ανησυχητικά μηνύματα σε ό,τι αφορά το έλλειμμα εμπορίου που έχουμε με το Βιετνάμ και μα προειδοποιούν ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα μετά την επικύρωση. Στέκει αυτό. Και τι προσδοκίες έχουμε στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα οι σκιώδει εισηγητέ από πλευρά του ΕΛΚ, ο κύριο Βίνκλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις πολύ χρήσιμες, για τις πολύ χρήσιμες ε, παρουσιάσεις από τη, την Ομοσπονδία των Συνδικάτων, από τον ΠΟΕ. Σας ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες αυτές που μας δώσατε. Νομίζω από πλευράς του ΕΛΚ διαπιστώνουμε μια πολύ καλή αξιολόγηση και επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Μιλτήριο. Από πλευρέ του ΕΛΚ, λοιπόν, και εμεί προσπαθούμε να διακρίνουμε αυτού του σημαντικού πυλώνε, αυτέ τι βασικέ γραμμέ. Οικονομικό αντίκτυπο, προώθηση των αλλαγών στην κοινωνία, γιατί θέλουμε να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες και να προωθήσουμε λοιπόν τέτοιες ε, αλλαγέ μέσω των ευρωπαϊκών, μέσω τη νέα συμφωνία και κατά τρίτον τα γεωπολιτικά ζητήματα. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Είναι η δεύτερη ημέρα που δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υποτίθεται ότι θα είναι γεωπολιτική στο χαρακτήρα τη. Δεν ξέρω αν θα είμαστε κι εμεί γεωπολιτικό κοινοβούλιο. Θα φανεί αυτό στην πορεία, αλλά είμαι βέβαιο ότι πολλά γεωπολιτικά ζητήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο της συζήτηση εδώ στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, γιατί το Διεθνές Εμπόριο είναι το μέσο το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να παρέμβουμε σε αυτά τα πολύ περίπλοκα ζητήματα. Τρεις σύντομες λοιπόν ερωτήσεις. Καταρχάς προς ε, το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο, Εμπορικό Επιμελητήριο. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα του κατά πόσον αυτή η νέα συμφωνία ηλεκτροεμπορίου θα επιφέρει αλλαγές. Τι δυναμικό υπάρχει εδώ και τι δυνατότητα υπάρχει σε ό,τι αφορά το Βιετνάμ. Πιστεύετε ότι ανταπεξερχέστε στις κοινωνικέ σα ευθύνε και στο Βιετνάμ. Φυσικά έχετε ευκαιρίες σε επιχειρησιακό, επιχειρηματικό επίπεδο. Αναλαμβάνετε όμω και την κοινωνική σα ευθύνη στο Βιετνάμ. Αυτή είναι η ερώτηση. Στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Εντυπωσιάστηκα. Εντυπωσιάστηκα για τις παρατηρήσεις σας, για την φιλοσοφική φύση και ο κύριος Λί νομίζω ότι το έθεσε το θέμα αυτό. Είναι φιλοσοφικό το ζήτημα σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα του σοσιαλιστικού συστήματος και τη ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση στο μέλλον. Είναι σαφές. Αλλά ασφαλώς ε, είναι και δύσκολο περιβάλλον το Βιετνάμ. Πριν από μόλι τέσσερι δεκαετίε αν το σκεφτούμε, αντιμετώπιζαν προβλήματα περιβαλλοντικά μετά τον πόλεμο και το θέμα των ατόμων με αναπηρία. Σημαντικό ζήτημα ακόμη και σήμερα. Ερωτώ λοιπόν, Επίσης, κύριε Λί, αναφέρατε το περιβάλλον της Νοτιού Κορέα, της Ιαπωνίας, της Σιγκαπούρης. Πιστεύετε ότι το Βιετνάμ θα μπορούσε να αποτελέσει μια κινητήριο δύναμη για να προωθήσει τα εργασιακά δικαιώματα και κυρίως και τη στάση έναντι των συμβάσεων του ΠΟΕ. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σύντομη ερώτηση για να συμφωνήσω και με τον εισηγητή που έθεσε επίσης το ερώτημα αυτό. να ρωτήσω πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε. Γιατί αναφέρουμε τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από την Κίνα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Κερντάλινγκ. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Πραγματικά ήταν πολύ πλούσιες αυτές οι παρουσιάσεις και νομίζω ότι ε, πολλές ερωτήσεις ε, προέκυψαν από πλευρά μα. Ε, είναι σαφέ ότι η μεταρρύθμιση του εργασιακού κωδικά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό. Και αυτό αποτέλεσε μεγάλο κομμάτι τη επίσκεψη στο Χανόη τέλη Οκτωβρίου. Να τονιστεί ακριβώ η σημασία τη αλλαγή αυτή και ε, να τονίσουμε και ότι είναι σωστό δρόμο αυτό. Να πω ευθύ εξ αρχή αυτό που σχολίασε ο κύριος Λί σε ό,τι αφορά την ισχυρή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΟΕ των ε, Υπουργείων στο Βιετνάμ και άλλων φορέων στο εξωτερικό για να δημιουργηθεί τελικά ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την επικύρωση των συμβάσεων του ΠΟΕ και τη μεταρρύθμιση του εργασιακού κώδικα. Ε, χρειάζεται λοιπόν ένα δίκτυο υποστήριξης. Ε, θέλουμε επίσης και τεχνική αρρωγή από την άλλη πλευρά ε, να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Να κάνω και εγώ τρεις ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Μία ερώτηση καταρχάς ε, προ την ε, Eurochambers. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για σειρά ετών, εξετάζουμε το θέμα του κεφαλαίου και του βιώσιμη ανάπτυξη σε ό,τι αφορά το εμπόριο και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή τους. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν την άποψη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μια τέτοια χώρα τι πιστεύετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε για να μπορεί να είναι πιο εφαρμόσιμες αυτές οι διατάξεις του κεφαλαίου εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το Μάιο φέτος η Βιντιναμέζικη Συνέλευση έκανε μια πολύ έντονη συζήτηση για την ε, χρήση του ποινικού κώδικα σε ό,τι αφορά την καταναγκαστική εργασία στι ιδιωτικέ επιχειρήσει στο Βιετνάμ. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να ακούσουμε οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει τι πίστευαν και τι έλεγαν στην όλη αυτή η συζήτηση όταν ε, εθίχθησε το θέμα αυτό της καταναγκαστικής εργασίας στο Βιετνάμ. Κατά πόσον υπήρξε σωστή εκπροσώπηση, κατά πόσον υπήρχαν ευρωπαϊκές χώρες και επιχειρήσεις οι οποίες να τοποθετήθηκαν στην όλη συζήτηση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να το, ξέρουμε αυτό. Γιατί προφανώς αυτό συνάδεκε με τη συνθήκη υπαριθμών 105. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε προ τον ΠΟΕ. Να επανέλθω στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΟΕ και Βιατναμεζικών Αρχών. Στου κόλπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζουμε το πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μέσω της διαδικασία επικύρωσης να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία έτσι περαιτέρω. Προφανώ εδώ υπάρχει ένα περιθώριο μόχλαυση μέχρι ότου να γίνει η ψηφοφορία για την επικύρωση στι αρχέ του επόμενου έτου, κατά πάσα πιθανότητα. Εκεί μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή. Μία ιδέα όμω είναι να υπάρχει ένα κοινό, αξιόπιστο και σωστό οδικό χάρτη για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως και η επικύρωση τη ε, συνθήκη. Τι θα συμπεριλαμβάνονταν λοιπόν στον δικό χάρτη αυτό, πώς τον πλασιώναμε και θα μπορούσατε, θα θέλετε να συμμετέχετε για να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της συνεργασίας αυτής. Και η τελευταία ερώτηση προς ε, την Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Τονίσατε πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση μεταξύ των συνδικάτων, της ελευθερίας του συνδικαλίστησα και των ε, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Είπατε ότι υπάρχει μία ανησυχία σε ό,τι αφορά την καταπίεση των ε, αμοιβών, σε ό,τι αφορά τι συλλογικέ συμβάσει σε εργασιακό επίπεδο. Προφανώ. αν υπάρχει κατακαιρματισμό των αντιπροσώπων των εργαζομένων και αν δεν υπάρχει δυνατότητα ε, τομεακή εθνική οργάνωση ε, των εργαζομένων, τα ξέρουμε όλα από την ιστορία των συνδικάτων μα. Ε, αποτελούν θέματα όλα αυτά τα θέματα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, θεωρεί ο ΕΤΟΚ, για να μην υπάρξει αυτό ο αρνητικό αντίκτυπο στου εργαζόμενου εργαζόμενους του Βιετνάμ και να υπάρχει θετικό αντικτύπο σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και, κατε... το ξατεξίνη. Ευχαριστώ πολύ. Τρινιού τώρα, η κυρία Κάλτσπρο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ε, Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σας ευχαριστώ για την επίσκεψή μας στο Βιετνάμ. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα και ήταν ε, πολύ χρήσιμο να πάμε στο νέο ακριβώ ε, πριν από τις αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε. Βλέπουμε ότι το εμπόριο είναι κάτι που όλοι το γνωρίζουμε καλά, έχουμε εμπορικές συμφωνίες, αυτό αποτελεί έναν τρόπο ε, συνεργασίας έτσι ώστε να έχουμε κοινή βούληση, κοινέ προϋποθέσεις, ακόμη και αν οι αρχικές θέσεις είναι διαφορετικές. Θέλουμε να είναι δίκαιο το εμπόριο, αλλά και να μπορεί να ευνοεί την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ευημερία στις διάφορες χώρες. Επίσης, το εμπόριο αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό βιωσιμότητας. Σήμερα έχουμε ξεκάθαρα κεφάλαια για το τι πρέπει να κάνουμε, επί των οποίων πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη γνωμοδότηση. Σε ό,τι αφορά το κλίμα έχουμε και τη Συμφωνία των Παρισίων και μπορούμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την κλιματική συμφωνία. Όμως η βιωσιμότητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όλων, όλου αυτού του μηχανισμού. Και υπάρχει και στη συμφωνία με το Βιετνάμ και πραγματικά είναι πολύ καλό που ακούμε ότι υπάρχουν θετικά μηνύματα από το Βιετνάμ ε, σε σχέση με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνδικαλιστικές σχέσεις, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική βιωσιμότητα στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά αυτή την κοινωνική βιωσιμότητα, είναι προφανές ότι πρέπει να βασιστούμε και σε ένα πλαίσιο ελευθερίας έκφρασης, να υπάρχει δυνατότητα να μπορεί ο καθένας να εκφράσει τη βούλησή του και από κοινού να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να υπηρεσπίσουμε τα σημαντικά για μας θέματα. Αυτές είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Ε, είπαμε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος, σημαντικά μηνύματα που εστάλησαν την περασμένη εβδομάδα ε, και ε, ελήφθησαν αποφάσεις ε, στην Εθνοσυνέλευση, όμω ε, ταυτόχρονα είδαμε και κάποια σοκαριστικά μηνύματα που έδειξαν ότι η κατάσταση ό,τι φορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών διακυβεύεται. Είχαμε τη σύλληψη κάποιων blogger. Αυτά μας προκάλεσαν κάποιες αμφιβολίες. Λοιπόν, έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το ρόλο που μπορούμε εμείς να διαδραματίσουμε σε ό,τι αφορά το Βιετνάμ να σεβαστεί τις υποσχέσεις του στα εργασιακά. Γιατί είναι προφανές ότι εδώ πρόκειται για θέματα που θα πρέπει να αποκρισταλωθούν στην νομοθεσία. Αλλά φυσικά αυτό το θέμα ενδιαφέρει τους πάντες. Όλοι θα πρέπει να βελτιώσουν τις ε, υφιστάμενες δυνατότητες για να μπορέσουμε να έχουμε πιο στενές ε, σχέσεις. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στον λόγο τομέα και κάτι ακόμα. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα της ελευθερίας έκφρασης και της δυνατότητα να μπορεί κάποιος να κάνει τη φωνή του να ακουστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους εργοδότες αλλά και για τα συνδικάτα. γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική και λειτουργική οικονομική ζωή. Και θα ήθελα να μου πείτε και τη γνώμη σας για τον κοινό δικό χάρτη. Δηλαδή να δούμε τι follow-up μπορεί να υπάρξει και σε αυτή τη συμφωνία. Γιατί έχουμε τεράστιες δυνατότητες που δίνονται στην οικονομική ανάπτυξη και για να έχουμε και ένα πιο βιώσιμο κόσμο. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε τα θέματα αυτά και τι πιστεύετε για την δική σας συνεισφορά. Πώς μπορείτε εσείς να συνεισφέρετε. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω στα γαλλικά. Ζητώ συγγνώμη, σα γυρνάω την πλάτη, αλλά πρέπει η φωνή μου να φτάνει στο μικρόφωνο για να μπορώ να με μεταφράσουν. Θα ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις που απευθύνονται στο εμπορικό επιμελητήριο. Μιλήσατε για ένα γεωστρατηγικό σημαντικό θέμα. Μπορώ να καταλάβω τι λέτε για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το Βιετνάμ. Επίσης αναφέρεστε και στο ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη του περιφερειακού ανταγωνισμού. Θα ήθελα όμως να πω σε σχέση με αυτό που είπατε όσον αφορά τις θετικές επιπτώσεις και ακριβώς επειδή μιλήσαμε και για το εμπορικό έλλειμμα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει, εκτός και αν υπάρχουν κάποιες νέες πληροφορίες που δεν γνωρίζουμε. Το θέμα επίσης του due diligence που αφορά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ποια είναι η δέσμευση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όσον αφορά τις μελλοντικές επενδύσεις, αλλά και αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και των παιδιών ειδικότερα. Μιλήσατε για καλύτερους μηχανισμούς ε, για την επίλυση των διαφορών, κάτι που θα βοηθήσουν να αυξηθούν οι επενδύσεις από το εξωτερικό. Τι σας επιτρέπει να πείτε κάτι τέτοιο, έχετε επιχειρήματα ιδιαίτερα για το Βιετνάμ. Τέλος, Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, αυτό είναι απαραίτητο να γίνει πριν την ύπαρξη συμφωνίας. Όλοι ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι συμφωνίες και να υπογράψουμε, ό,τι και να γίνει στα πλαίσια του, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, δεν υπάρχει περίπτωση να τηρηθούν και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σε σχέση με τον ε, ποινικό κώδικα, λοιπόν, μήπως κάναμε τα πράγματα ανάποδα. Διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει και δεν διασφαλίζεται η ελευθερία του συνεταιρίζεστε, πώς ε, μπορούμε να μιλάμε για υπογραφή νέων συμφωνιών. Πριν από λίγα χρόνια ήταν αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι το Βιετνάμ θα σεβόταν αυτές τις ελευθερίες. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και τα ανεξάρτητα συνδικαλιστικά όργανα, τους ανεξάρτητους φορείς, γιατί πολλές φορές παρουσιάζουν διαφορετικά την κατάσταση. Μιλήσατε για τους τομείς, τις επιχειρήσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει εγγύηση και σεβασμός όλων αυτών των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σε όλους τους τομείς. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω όσον αφορά τα πιο ενημερωμένα στοιχεία, τα πιο πρόσφατα στοιχεία που να μας δείχνουν ότι μειώνεται η εργασία των παιδιών. Τέλος, για την τελευταία παρέμβαση θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτά που αναφέρατε. Τα πιο πολλά δηλαδή ερωτήματα που θέσατε είναι και ερωτήματα των πρασίνων. Ιδιαίτερα ότι πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση και ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Σήμερα εγώ δεν θεωρώ ότι ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας αυτών των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και την ε, προστασία θεμελιωδών αρχών όπως η ελευθερία έκφρασης. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις και την ίδια ώρα συλλήψεις πολιτικών κρατουμένων. Μάλιστα αναφερθήκαμε σε μία από αυτές. Θα πρέπει πραγματικά η κυβέρνηση του Βιετνάμ να δείξει αποφασιστικότητα για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, πριν εμείς περάσουμε στην επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης. Με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα το χρονοδιάγραμμα, αν υπάρχει ο δικός χάρτης. Αυτό είναι μια θέση πάγια των πρασίνων. Πρόκειται για ένα βήμα σε μια διαδικασία που θα πρέπει να συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε χρόνο. Η Επιτροπή μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα, είναι διατηθμένο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις μαζί σας, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο. Πρόεδρος, ο Σκαναλτίνη δεν είναι παρόν. Θα πάρω εγώ το λόγο για το ID. Βεβαίω και είμαστε υπέρ μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε για την Ευρώπη αλλά και για το Βιετνάμ. Πρόκειται για μια περιοχή, η Νότια Ανατολική Ασία, που αναπτύσσεται με τους ε, βαθμούς ανάπτυξης. Ε, η οικονομική ανάπτυξη σίγουρα θα δημιουργήσει και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και περισσότερη ελευθερία στους πολίτες. Ακριβώς λοιπόν επειδή εξετάζουμε συνήθως αυτές τις εμπορικές συμφωνίες όσον αφορά τις οικονομικές τους επιπτώσεις και όχι τις πολιτικές τους επιπτώσεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις παρόλα αυτά. Υπάρχουν εγγύησεις για τα πνευματικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που επενδύουν στο Βιετνάμ. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα από τα πιο εμφανή προβλήματα που παρουσιάζονται όταν ε, δραστηριοποιούμαστε στην Κίνα. Τι μπορείτε να μας πείτε για την κατάσταση στο Βιετνάμ και αν αυτή πραγματικά διαφέρει από αυτό που συμβαίνει στην Κίνα. Επίσης, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες όσον αφορά την προστασία των ε, ξένων επενδύσεων στη χώρα σας. Πώς μπορούμε επίσης να βγάλουμε τα κέρδη των επιχειρήσεων από το Βιετνάμ. Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις μεταφορές ποσών κεφαλαίων που αφορούν τις ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις από το Βιετνάμ. Πώς μπορούν οι επενδυτές, οι ευρωπαίοι επενδυτές να μεταφέρουν τα χρήματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Εμμανουέλ Ωραία από την ΚΟΥ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο συγγνώμη, και εγώ σας γυρνάω την πλάτη, αλλά είναι καλύτερα για να ακούγεται η φωνή μας. Ο κύριος Βίνκλερ είπε ότι πρόκειται για μια γεωστρατηγική συμφωνία. Έχει δίκιο. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Πρώτον, όσον αφορά το εμπορικό επιμελητήριο. Ναι, υπάρχουν εντυπωσιακοί ρυθμοί, η ανάπτυξη στο Βιετνάμ είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για ένα νέο εργαστήριο που ουσιαστικά εντυπωσιάζει και προσελκύει πολλούς Ευρωπαίους επενδυτές. Ο εισηγητής μας είναι πολύ ειλικρινής, το κείμενό του αναφέρει ότι είναι ανταγωνιστική χώρα το Βιετνάμ γιατί έχει πολύ χαμηλά ε, επίπεδα μισθών, αποδοχών των εργαζομένων. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Όμως αν κοιτάξει κανείς ε, το έλλειμμα, το 2008 ήταν 5 εκατομμύρια και περάσαμε σήμερα στα 30 εκατομμύρια. Έλλειμμα το οποίο θα γίνει 40 εκατομμύρια. Μα αν κοιτάξει κανείς αυτή την τάση, διαπιστώνει ότι δεν είναι win-win αυτή η κατάσταση. Δεν ε, είναι από τις δύο πλευρές τα ωφέλη. Διαπιστώνουμε ότι στην κλωστοεφαντουργία, παραδείγματο χάρη, έχουμε δύο εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένος κίνδυνος, όχι μόνο στον τομέα της κλωστοεφαντουργίας, αλλά και σε άλλους τομείς, να πληγεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από αυτές τις σχέσεις με το Βιετνάμ. Τέλος, το θέμα της μη διάκρισης, της διαφάνειας, της πρόσβασης σε πολλές αγορές, τη δυνατότητα δίσδυσης σε κάποιες αγορές μέσω υποβολής προσφορών. Διαπιστώνω ότι τα εμπόδια μειώνονται σταδιακά, αλλά με πάρα πολύ χμηλούς Βλέπουμε τα 40 δισεκατομμύρια που είναι το ανώτοτο κατόπλη αυτή τη στιγμή, πώς μπορούν οι επιχειρήσεις μας, αν θέλετε, να διεισδύσουν σε αυτή την αγορά. Γιατί εκτός από τους μεγάλους ομίλους δεν βλέπω τον τρόπο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, να υποφεληθούν από αυτή τη συμφωνία. Δεν κατάλαβα και πολύ καλά βέβαια τι είπατε, γιατί εγώ βλέπω την έκθεση που λέει ότι η σύμβαση του 87 θα αρχίσει να ισχύει το 20 ή το 21. Τι ακριβώς ισχύει. Είναι κάπως αντιφατικά αυτά που ακούμε. Ακούμε για την ελευθερία των συνδικαλιστικών οργανώσεων το 21 ή το 23. Αν κατάλαβα καλά, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις, αυτό θα ισχύει από τώρα. Κατάλαβα καλά ότι οι νέες διατάξεις που απορρέουν από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα γίνονται μέσω του επίσημου συνδικαλιστικού οργάνου. Και όλες οι ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν θα μπορούν να διαπραγματευτούν και πολλά πράγματα. Αυτό βέβαια είναι μια ερώτηση για την ΔΟΕ. Μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, αλλά θα συμφωνήσω με την προηγούμενη ομιλήτρια ότι ό,τι και να συζητάμε όσον αφορά τις συλλογικέ συμβάσεις και διαπραγματεύσεις, εάν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, από τη στιγμή δηλαδή που είναι ποινικό αδίκημα η επίκριση ε, της κυβερνητικής πολιτικής, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει περισσότερη ελευθερία. Όπως ξέρετε, τιμωρείται σήμερα η προπαγάνδα κατά του σοσιαλιστικού κράτους του Βιετνάμ. Η απεργία αποτελεί τμήμα προπαγάνδας. Όλες επίσης αυτές οι διατάξεις που προβλέπουν ε, κυρώσεις για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Τις ε, προσπάθειες και τα σχέδια της κυβέρνησης του Βιετνάμ τι ακριβώς εννοούν αυτές οι, αυτή η συγκεκριμένη διατύπωση αυτών των διατάξεων. Ναι, υπάρχει πρόοδος, όμως στην πράξη η νομοθεσία δεν βλέπω να μεταρρυθμίζεται και να αλλάζει όταν ποινικοποιείται η απεργία, παραδείγματο χάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στο θέμα της ανησυχίας της εφαρμογής. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή του εξής. Ποιες προοπτικές υπάρχουν ε, προκειμένου το Βιετνάμ να θετήσει τις κατάλληλες διατάξεις ε, για να διασφαλίσει ότι όλες οι δεσμεύσεις ε, σε ό,τι φορά το εργατικό δίκαιο θα υλοποιηθούν ε, ακούσαμε την, τον εκπρόσωπο ε, της Διεθνούς Νομοσπονδίας Συνδικάτων αναφέρθηκε στην ε, δυσκολία ε, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες οργανώσεις. Επίσης αναφερθήκατε στη δυσκολία να συνδυαστεί το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε με το δικαίωμα του ελεύθερου συνδικαλισμού. Πώς το βλέπει αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, θα ήθελα να μάθω το εξής. Έχουμε κάποιες ανησυχητικές πληροφορίες σε σχέση με την ομοθεσία της ε, διαβίβασης δεδομένων ε, και της προστασίας της ιδιωτικότητας. Πώς είναι η κατάσταση αυτή και πώς θα εγγυθούμε ότι θα γίνονται σεβαστές οι αρχές που διέπουν αυτά τα δικαιώματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Τέλος, ε, ο δικός χάρτης, ο συγκεκριμένος προγραμματισμός για να μπορέσουμε να εγγυθούμε ότι θα υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις. Θα υπάρξει συμμετοχή και των ε, οργανώσεων και των εξωπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στην εκπόνηση του χάρτη πορείας και στην ανάπτυξή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη ΔΟΕ. Κύριε Λί, να ρωτήσω κι εγώ κάποια πράγματα. Έγινε μεγάλη συζήτηση για το θέμα της, ε, εφαρμοστής, της εφαρμογής της συμφωνίας ε, και της επικύρωσης ε, των δύο εκκρεμών συμβάσεων της ΔΟΕ. Αν κάνατε ένα σύντομο κατάλογο των πιο σημαντικών βημάτων για την εφαρμογή, ποια θα ήταν τα τρία, οι τρεις πιο σημαντικές δράσεις που θα έπρεπε να αναλυφθούν για την εφαρμογή και της Συμφωνίας και των Τριών Συμβάσεων ΔΟΕ και στην Κομισιόν να θέσω το εξή ερώτημα. Επίσης, ακούσαμε από τα συνδικάτα ότι είναι απαραίτητη οικοδόμηση ικανοτήτων. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε την οικοδόμηση ικανοτήτων μαζί με τη ΔΟΕ και τι πόρους έχει στη διάθεσή της η Κομισιόν για την οικοδόμηση ικανοτήτων στο Βιετνάμ. Και ποιε είναι οι σκέψεις σας ε, για το πώς θα υποστηρίξετε την οικοδόμηση ικανοτήτων ε, υπό το φως της εφαρμογής ε, των συμβάσεων εδώ στο Βιετνάμ. Και για να ξεκινήσουμε με διαφορετική σειρά τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Ευχαριστώ. Στο θέμα της εμπίεσης των μισθών και το τι να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε τα νομοθετικά μέσα που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή του δικαίου και να διασφαλίσουμε ότι ε, με την εγγραφή των θα υπάρξει ικανότητα συνεργασίας ε, για να ε, μπορέσουν ε, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα βάσει συλλογικών διαπραγματεύσεων από κοινού, όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων. Δηλαδή, όταν κάνεις αυτή τη μείωση, θα πρέπει να μπορέσεις να διασφαλίσεις ε, ότι υπάρχει και ο χώρο να συμμετέχουν οι οργανώσεις εκπροσώπων των εργαζομένων. Θα πρέπει να υπάρξει κοινή διαπραγμάτευση, προκειμένου να καθοριστούν και μισθοί που θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί καθορισμού των μισθών. Δηλαδή, για να καθοριστεί πώς ε, θα γίνει, πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις για του μισθούς. Γιατί ε, μπορεί να έχεις διαφορετικές ε, φόρμουλες, παραδείγματος χάρη, για τον καθορισμό των μισθών. Και αυτό θα αποδυναμώσει περαιτέρω τα συνδικάτε, μάλλον την διαπραγματευτική διαδικασία και δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρειάζεσαι λοιπόν οικοδόμηση ικανοτήτων. Έτσι λοιπόν, εργανώσει εκπροσωπών εργαζομένων, τα συνδικάτα, όποιο και αν ε, συμμετέχει σε διαπραγματεύσει πρέπει να έχουν τι σχετικέ ικανότητε. Ε, και γι' αυτό και η Συνομοσπονδία Συνδικάτων βλέπει να υπάρχει κάποιος ε, ρόλος στο να εργαστούμε με τις οργανώσεις εκπροσωπών εργαζομένων αλλά και ανεξάρτητες οργανώσεις που θα ανακύψουν από τη διαδικασία. Έτσι απαντούμε στο θέμα αυτό. Και να προσθέσω ότι ο ίδιος ο μηχανισμός για τον ελάχιστο μισθό θα πρέπει να ακολουθηθεί ως παράδειγμα. Και αν δεν είναι ισχυρός θα πρέπει να βοηθηθεί, θα πρέπει να υποστηριχθεί προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κατάλληλοι μηχανισμοί και φόρμουλες υπάρχει για υπάρχουν για τον καθορισμό των μισθών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ εκπρόσωπο τη ΔΟΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, για την συμβουλευτική ομάδα. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, διαφορετικές εκτιμήσεις για την συμβουλευτική ομάδα σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά στο πλαίσιο του Βιετνάμ βλέπω ότι υπάρχει ένα εμπόδιο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημόσιος χώρος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή για ΜΚΟ για να υπάρξει διάλογος με την κυβέρνηση σε ισότιμο επίπεδο. Και αν συσταθεί αυτή η συμβουλευτική ομάδα θα είναι το πρώτο φόρουμ όπου οι ΜΚΟ σε περιβαλλοντικό και εργασιακό επίπεδο θα μπορούσαν να θέσουν τις απόψεις τους στην κυβέρνηση. Έτσι βλέπω την πιθανή συνεισφορά αυτής ε, της συμβουλευτικής ομάδας. Η κυβέρνηση αρχίζει να δίνει προσοχή τώρα σε αυτή την εγχώρια συμβουλευτική ομάδα και συζητούν τώρα ποια θα είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διορίσουν τις ΜΚΟ που θα συμμετέχουν στη συμβουλευτική ομάδα. Ελπίζω τα κριτήρια να είναι δίκαια και δημοκρατικά και διαφανή. Όμως κατά τα δεν έχει ληφθεί κάποια άλλη δράση, επομένω δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω. Δεύτερον, για την ε, συμβατότητα τώρα του συσχετιστικού στήματο και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε Το πολιτικό γραφείο της ε, Βιτναμιζική κυβέρνησης ε, έθεσε το θέμα αυτό και μάλιστα ε, ρωτήθηκε ο Υπουργός ε, Εργασίας και δεν ήξερε πώς να απαντήσει. Και εγώ έγραψα για το πώς μπορεί να είναι συμβατά αυτά και κατόπιν το πολιτικό γραφείο έδωσε το πράσινο φως. Ναι, μπορείτε να προχωρήσετε και τώρα είμαστε πεπισμένοι ότι είναι συμβατό. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και τα σχετικά έγγραφα. Όμως ε, θέλω να διευκρινίσω σε αυτό το πλαίσιο το γεγονός ότι το Βιετνάμ έχει θετήσει τον εργατικό κώδικα που ε, συμπεριλαμβάνει ισχυρό στοιχείο του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε σημαίνει ότι το Βιετνάμ αρχίζει να ακολουθεί από μια διαφορετική οδό από την Κίνα και υπήρχε ήδη αυτό. Είχαμε διάκριση μεταξύ εκτελεστικού και νομοθετικού σώματος ε, αλλά και με την υιοθέτηση του εργατικού κώδικα το Βιετνάμ ακολουθεί τη δική του οδό και νομίζω ότι πρέπει να την ενθαρρύνουμε στο θέμα του δικού χάρτη. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ το θέμα του δικού χάρτη, αλλά σας πω δύο ιστορίες. Ε, την ημέρα της υιοθέτηση του εργατικού κώδικα ε, ε, είπε ο κύριος είπα στον κύριο εμπνευστή ότι πρέπει να το γιορτάσουμε με κρασί. Όμως μου είπε ότι δεν είχε χρόνο γιατί ήταν σε μια επιτροπή και συζητούσε ένα πιθανό εμπόδιο για την κύρωση της σύμβασης 105 και έπρεπε να μείνει μέχρι τις 10 το βράδυ για να άρει το εμπόδιο αυτό. Δηλαδή, ακόμη και εκείνη τη μέρα είχε υιοθετηθεί το εργατικό, ε, ο εργατικός κώδικας, ε, δούλευε η υπεύθυνη για την υιοθέτηση της Σύμβασης 105. Και αύριο, να σας πω δεύτερη ιστορία, πρέπει να πάω στο Ανόη για να συμμετέχω σε μια συνάντηση των Υπουργείων για την εφαρμογή του εργατικού κώδικα. Λαμβάνουν λοιπόν δράση. Υπήρχε μια ερώτηση για το πώς θα αναπτυχθεί ο ειδικό χάρτης, νομίζω. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο του. Γιατί, όπως είπα, ποια είναι, τι διαφοροποιεί το Βιετνάμ από την Ιαπωνία, πριν το σχάρι Το θέμα είναι ο συντονισμό και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΔΟΕ ε, και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετναμιστικής Κυβέρνησης. Αυτό δεν το είχαμε στην περίπτωση της Κορέας, της Ιαπωνίας και της Σιγκαπούρης. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν καλύτερα αυτή τη φόρμουλα που λειτουργήσε έχουμε την απάντηση για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή τα όσων συμπεριλαμβάνονται στη ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και στο κεφάλαιο της ε, βιώσιμης ανάπτυξης και εμπορίου. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσω τις επόμενες μέρες και εβδομάδες με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνομιλούσαμε την πρεσβεία σα στο ΕΝΟΗ κάθε εβδομάδα. Δεν ισχύει αυτό για τι άλλε χώρε. Αυτό δημιούργησε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Δεν ε, έχει ολοκληρωθεί βέβαια η όλη διαδικασία. Κλείνουμε κεφάλαιο, προχωρούμε στο επόμενο. Εργαζόμαστε τώρα στην υιοθέτηση του εργατικού κώδικα. Σας ευχαριστώ κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ακούστηκαν σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που θα πρέπει να απαντήσει ακόμα η ΔΟΕ. Τα πιο βασικά στοιχεία για την εφαρμογή των τριών ε, βασικών ε, συμφωνιών του ΔΟΕ είναι το θέμα της νοτροπίας. Θεωρώ αυτό τα λέει καλύτερα από όλα. Δεδομένη της ρεαλιστικής αντιμετωπίσης ε, του Βιετνάμ, θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνουν πολλές από τις αλλαγές που χρειάζονται, αλλά το να αλλάξει το βαθύ κράτος, α, το αποκαλέσω έτσι, ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση, αυτό θα πάρει χρόνο. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά όμως, τρία βασικά θέματα θα πρέπει να ρυθμίσουμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, σε ό,τι αφορά την καταχώρηση των ανεξάρτητων συνδικάτων ή κατά δεύτερον η δυνατότητα των εργαζομένων να κάνουν διαπραγματεύσει για σωστέ συλλογικέ συμβάσει, γιατί η συλλογική σύμβαση αποτελεί και μια ικανότητα και κατά τρίτον σε η διευθέτηση των ζητημάτων, γιατί εδώ είναι καινούριο ο κλάδο αυτός. Κατέθεσε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα και πώ θεωρούμε ότι είναι η σχέση του με την επικύρωση τη σύμβαση για την 105, για παράδειγμα. Όταν ε, κοιτάμε την επικύρωση μιας συνθήκης, δεν κοιτάμε ε, απαραίτητα το θέμα της επικύρωσης και της καταχώρησης, γιατί η επικύρωση ε, γίνεται ένα χρόνο μετά την καταχώρηση. Κοιτάμε λοιπόν αυτή την διάμεση περίοδο τι γίνεται σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στον ποινικό κώδικα πρωτού καταχωριστεί η συνθήκη. Εδώ έχουμε να πούμε το εξή. Σε διάφορες περιπτώσεις, ακόμα και αν κυβερνήσεις κάνουν ε, βήματα τα οποία συνάδουν με τη συνθήκη, πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στη συνέχεια. Έχουμε κάποια γραπτά σχόλια σε ό,τι αφορά τις διατάξεις οι οποίες αναφέρονται. Πιστεύουμε ότι γενικά πολλές από τις διατάξεις του ποινικού κώδικα όντως δίνουν ε, μεγάλες, υπερβολικά μεγάλες ε, αρμοδιότητες στις κυβερνήσεις ε, προκειμένου να υπάρχει πολιτική αποτελεσματικότητα και αυτό θα συνεχιστεί με βεβαίως, ακόμα και μετά την επικύρωση. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για την παιδική εργασία, υποστηρίζουμε τις αρχές. Κάνουμε μία μελέτη για την παιδική εργασία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτά αναφέρθηκαν και στον οδικό χάρτη σε ό,τι αφορά το θέμα για τη σημαντική ε, μείωση των ε, περιστατικών καταναγκαστικής παιδικής εργασίας, σε ό,τι αφορά το θέμα της συμβατότητας με το σοσιαλιστικό σύστημα. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να στριχτούμε στην ε, ρεαλιστική αυτή η προοπτική. Φυσικά υπάρχουν θέματα σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα. Αλλά πιστεύουμε ότι τα ωφέλη τα οποία θα διακρίνουν οι αρχές και στην συμφωνία αυτή αλλά και σε άλλες συμφωνίες ελευθερειομπορίου θα τους οδηγήσουν να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία μεταρρύθμισης εν γέννη. Τώρα το Βιετνάμ αν θα καταστεί κινητήριο δύναμη για την επικύρωση και σε άλλα μέρη στην Νοτιοανατολική Ασία θεωρώ ότι είναι μάλλον απίθανο ότι το Βιετνάμ θα καταστεί ποτέ πρότυπο δεδομένης και της ιστορίας του ΑΣΕΑΝ και της μεγάλης ε, ποικιλία πολιτικών μοντέλων. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει, θεωρώ, την κινητήριο δύναμη. Αλλά παραν τούτου θεωρώ ότι το Βιετνάμ έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο και να, να δημιουργήσει πολύ να προκαλέσει μάλλον μεγάλη προσοχή από τις άλλες χώρες στην Ανατολική Ασία που είναι μάλλον απρόθυμες και θεωρώ ότι θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει κινητήριο δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Τσέμπερ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και χαίρομαι πολύ γιατί πολλέ από τι ερωτήσει αυτές ήταν εύστοχε. Χαίρομαι που έχω κάποια Δεύτερα, να απαντήσουμε, να τις απαντήσουμε μία προς μία και στην ερώτηση της ε, Σουηδίας, ε, αγγλικά και γαλλικά. Με τη σειρά, κύριε Βίνκλερ, αναφερθήκατε στις ε, συνέπειες οικονομικές και τις γεωπολιτικές. Όταν το TPIP και ο πρόεδρος ε, Τραμπ αποφάσισε να αποχωρήσει, ξαφνικά είδαμε ότι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά γκρεμίστηκε στο Βιετνάμ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε συναντήσεις με αξιωματούχους, με υπουργού, με τον Πρωθυπουργό, ε, μας δέχονται στο Βιετνάμ και είναι πολύ πιο εύκολο για μας σε σχέση πλέον με τις συναντήσεις που έχουν με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Βλέπουμε ότι έχει ενισχυθεί λοιπόν η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά το 1993 με το πρώτο μου ταξίδι στο Βιετνάμ υπήρχαν επενδυτές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία. Πέρσι μετά από 30 χρόνια άμεσων επενδύσεων δεν αναφέρθηκε τίποτα για τον ρόλο που παίζουν ε, οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις, τις μεγάλες επιχειρήσεις που έγινε, ε, και επενδύσεις που έγιναν το 1993. Αναφέρθηκε κάτι για τις επενδύσεις στη, από το Βέλγιο, από μια βελγική εταιρεία. Όμως πλέον τον κυριαρχικό και τον πρωταρχικό ρόλο παίζουν η Κορέα, η Κίνα και όλες οι ασιατικές χώρες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή της Ευρώπης σαν μία φωνή στο Βιετνάμ. Και βεβαίως εδώ το θέμα των μεταρρυθμίσεων, η δύναμη που μπορούν να, να ε, οι δυνάμεις που μπορούν να κινητοποιήσουν όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις αυτές οι επενδύσεις και το θέμα των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να συναντάμε τους υπουργούς, τους ηθήνοντες. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο. Αλλά έχουμε ξεκινήσει το 87, το 87 όταν ξεκίνησε αυτή η πρώτη προσπάθεια ε, επενδύσεων. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ελεύθερες συναλλαγές, δεν υπήρχε άνοιγμα στο Βιετνάμ για καμία ε, τέτοιου είδους εμπορική διαδικασία δραστηριότητα. Μετά από 30 χρόνια βλέπουμε ότι με τον τρόπο τους, που είναι ένας ε, αργός τρόπος και με τους αργούς ρυθμούς τους, Σιγά σιγά οι επιχειρήσεις κατάφεραν να αλλάξουν την κατάσταση. Έχουμε πλέον το φόρουμ μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και του Βιετάμ και σιγά σιγά οι μεταρρυθμίσεις ε, κερδίζουν ε, έδαφος. Πολλές φορές, επαναλαμβάνω, ο χρόνος ε, είναι ο κύριος αντίπαλός μας. Πολλές φορές μετά από τρία-τέσσερα χρόνια βλέπουμε μετά από συνεχείς επαφές και προσπάθειες να αλλάζει κάτι στην νομοθεσία. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι όλη η αγορά και όλες οι επιχειρήσεις ε, του Βιετνάμ είναι έτοιμες ε, για ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές. Όχι, αλλά κάποιοι τομείς έχουν ανοίξει, κάποιοι τομείς πλέον έχουν προχωρήσει. Τώρα, βεβαίως και είμαστε επιχειρηματίες, βεβαίως και έχουμε μια τεχνητή στήριξη, αλλά δεν είμαστε εμείς οι εμπειρογνώμονες. Γι' αυτό και προσπαθούμε να εξηγήσουμε στις αρχές του Βιετνάμ ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, πρέπει να γίνει πιο φιλική προς επενδύσεις. Βλέπετε εδώ σε αυτό το έντυπο για το 2019 όλες τις νεότερες εξελίξεις. Για το θέμα του περιβάλλοντος έχουμε πάρα πολλές συναντήσεις, πάρα πολλά συνέδρια, πάρα πολλές ομιλίες ε, για τη ε, περιβαλλοντολογική πολιτική. Και βεβαίως ε, το Βιετνάμ έχει υπογράψει τη συμφωνία του Θέλουμε να εξηγήσουμε στο Βιετνάμ ποιες είναι οι θετικές ε, επιπτώσεις από τη χρήση πράσινων ε, εναλλακτικών ε, τεχνολογιών, της ενέργειας, το θέμα του πλαστικού. Εξηγούμε στο Βιετνάμ ότι πρέπει το πλαστικό σιγά σιγά να αντικατασταθεί, όπως γίνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από άλλες ε, μορφές συσκευασίας. Αλλά όλα αυτά θα πάρουν χρόνο. Και βεβαίως ε, δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να γίνουμε μία κοινωνία, ούτε εμείς ούτε το Βιετνάμ που θα σεβόμαστε όλες τις αρχές και όλα ε, τα, όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Όλα όμως τα μέλη της, ε, των επιχειρήσεων από το Βιετνάμ που συμμετέχουν στο Ευρωβιετναμέζικο Εμπορικό Επιμελητήριο τηρούν τις ευρωπαϊκές αρχές. Υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές για την κατάρτιση των εργαζομένων και ήδη έχει ξεκινήσει μια πραγματική σύγκληση μεταξύ των μελών από το Βιετνάμ και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πολλοί πήραν το λόγο και μίλησαν για τον ε, οδικό χάρτη. Όταν ξεκίνησαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή, οι οποίοι ήταν παρόντες, τους εξηγήσαμε το θέμα των ε, διαφορετικών ε, επιτροπών, 60 διαφορετικές επιτροπές. Εγώ είμαι νομικός ο ίδιος, αλλά πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλοί τομείς στους οποίους το νομοτοπικό έργο προχωρούσε, τους δίναμε τις πληροφορίες, τους ενημερώναμε και αυτό ξεκίνησε στην αρχή-αρχή των διαπραγματεύσεων. Σήμερα θέλουμε πραγματικά να περάσουμε στην υλοποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συνέλεγων. Και έγινε εξαιρετική ε, εργασία και πραγματικά όταν άρχισαν να ισχύουν οι αρχές του ΠΟΕ στο Βιετνάμ, ακριβώς επειδή υπάρχει κεντρική εξουσία στο Ανόη, αλλά υπάρχουν και 63 περιφέρειες Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι 63 περιφέρειες του Βιετνάμ και το πιο απομακρυσμένο μέρος του Βιετνάμ πρέπει να κατανοήσει, να καταλάβει ποια είναι τα άρθρα, ποιες είναι οι διατάξεις του ΠΟΕ που ισχύουν, που εφαρμόζονται. Αυτό παίρνει χρόνια, μας πήρε χρόνια. Έχουν συμφωνήσει και τώρα πλέον εφαρμόζεται κιόλας. Δεν θέλουμε λοιπόν να επαναλάβουμε το ίδιο με την ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Και όταν υπογράφηκε αυτή η συμφωνία, εγώ πραγματικά είπα σε όλους τους υπουργούς, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας, είπα σε όλους αυτή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Γι' αυτό και θέλουμε αυτή η συμφωνία μέσω του εμπορικού επιμελητήριου Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, Βιετνάμ, να υλοποιηθεί με ταχύτητα τους ρυθμούς. Θέλουμε λοιπόν εδώ, στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ανόη, σε εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, να σας πούμε ότι τα σημεία αυτά τα οποία θα πρέπει να μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να εξηγηθούν. Το θέμα των άμεσων επενδύσεων, το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το Βιετνάμ έχει υπογράψει όλες τις συμφωνίες ε, ελεύθερων ε, συναλλαγών, ελεύθερων, ελεύθερου εμπορίου. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το ίδιο με αυτό που αντιμετωπίζουμε στην Κίνα. Το πρόβλημα στο Βιετνάμ δεν είναι η υπογραφή, δεν είναι η βούληση συμμετοχής, είναι η υλοποίηση, η εφαρμογή. Επαναλαμβάνω, η εφαρμογή παίρνει χρόνο, πρέπει πρώτα να εγκριθεί η διάταξη, να εγκριθεί το νομικό κείμενο και κατόπιν να υλοποιηθεί να εφαρμοστεί πραγματικά. Το θέμα της ε, μεταφοράς ε, των κερδών δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε εδώ στις Βρυξέλλες και μιλήσαμε για αυτό το θέμα των άμεσων επενδύσεων. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λειτουργεί χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Τα κέρδη μπορεί να μεταφερθούν, να βγουν από τη χώρα και δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με το νόμισμα, ούτε με τη ρευστότητα της χώρας αυτής. Δεν άκουσα πολλές φορές, μου έχει τεθεί το ερώτημα, αλλά δεν άκουσα ποτέ να υπάρχει πρόβλημα με το θέμα αυτό. Το θέμα της ταχύτητας είναι κάτι που άκουσα σε μία ερώτηση, αλλά εγώ τα στοιχεία που διαθέτω είναι τελείως διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι το θέμα του ελλείμματος μεταξύ Βιετνάμ και Ευρώπης είναι αυτό που περιγράψατε. Ένα προς τρία είναι τα νούμερα που έχω εγώ και είναι ακριβώς το ίδιο έλλειμμα με αυτό που υπάρχει και με την Ιαπωνία και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες όταν θέλουν να εξάγουν το Βιετνάμ είναι τα ίδια. Τεχνικές ε, δυσκολίες και εμπόδια. Αλλά πιστεύω ότι χάρη στην ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ όλες αυτές οι δυσκολίες θα εξαλειφθούν. Βεβαίως, οι εξαγωγές ε, των ε, επιχειρήσεων του Βιετνάμ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες ε, τις προϋποθέσεις, σε όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και όλο και περισσότερες ευρω... ε, και επιχειρήσεις λειτουργούν βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Αυτό που περιμένουμε όμως είναι να αυξηθούν οι επενδύσεις, ε, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στο Βιετνάμ. Και όπως είπα και στην ομιλία μου, Υπάρχουν 26 διαφορετικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ Βιετνάμ και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πολλές από αυτές είναι εξαιρετικές, διότι παραδείγματο χάρη είναι εμπορικές και κατασκευαστικές, είναι συμφωνίες ε, μεταξύ της Γαλλίας, της ε, Μεγάλης Βρετανίας ή της Γερμανίας για την κατασκευή ε, ενός έργου μιας γέφυρας του Βιετνάμ. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συμφωνίες συνεπάγονται επενδύσεις. Η ερώτηση τώρα της προστασίας των επενδυτών και τι μπορεί κάποιος να κάνει αν υπάρχει πρόβλημα Μπορεί κάποιος να προσφύγει σε μας, μπορεί να προσφύγει στις αρχές. Όμως το πιο βασικό είναι να υπάρχουν κανονισμοί, να υπάρχουν νομικά κείμενα που να εγγυώνται την προστασία των δικαιωμάτων. Μιλήσατε για τα πολύ μεγάλα σχέδια επενδύσεων, όχι μόνο όμως οι διμερείς συμφωνίες και με την Ιαπωνία αλλά και με την Γαλλία ε, δεν συμπεριλαμβάνουν μόνο τεράστιες επιχειρήσεις ή μεγάλους ομίλους. Υπάρχουν και πολλές μικρομισές επιχειρήσεις που μέσω αυτής της ε, συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μπορούν να συμμετέχουν σε έργα και να επενδύσουν ε, στο Βιετνάμ. Όσον αφορά τώρα τις δημόσιες αγορές, τις κρατικές προμήθειες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, είδα ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μπορούν να συμμετέχουν πλέον. Επαναλαμβάνει ο συνάδελφος όμως ε, υπάρχει αυτό το έντυπο το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία για το 2019. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε πέντε λεπτά να σχολιάσετε. Πέντε λεπτά, Πρόεδρε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και πάλι και μου δίνετε το λόγο και που διοργανώσατε σημερινή, τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ λοιπόν, ε, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την ΤΟΕ για την παρουσίαση, για την πολύ καλή συνεργασία επίσης ε, που είχαμε. όχι μόνο στην Επιτροπή τη Νοσημπορία αλλά και σε άλλε επιτροπέ συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Για να σα εξηγήσω γιατί πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η FTA και η APA θα είναι επωφελή και για μα και για το Βιετνάμ. Και φυσικά κατανοούμε τα θέματα τα οποία ανησυχούν τον κόσμο και τα έχουμε συζητήσει και εδώ και σε άλλε επιτροπέ. Το βασικό λοιπόν θέμα εδώ είναι ποιο θα είναι ο αντίκτυπο. Ε, έχει ήδη σημειωθεί από τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου στο Βιετνάμ και τι είδου μόχλευση έχει υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεχιστεί αυτή η δέσμευση με το Βιετνάμ για να υποστηριχθεί η διαδικασία μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, τι ε, συμφωνίε αυτέ. Αποτελούν τον ιδανικό τρόπο. Η εφαρμογή ωστόσο θα είναι το βασικό στοιχείο. Πολλέ είναι οι διατάξει οι οποίε θα εφαρμοστούν μέσω τη ε, Σύμφωνη Ελευθερίου Εμπορίου. Κάποιε άλλε θα είναι μεταβατική, με κάποια μεταβατική περίοδο σε ό,τι αφορά τι προμήθειε, για παράδειγμα. Ανακοινώθηκε πρόσφατα πότε σκοπεύει το Βιετνάμ να επικυρώσει τι δύο υπόλοιπε συνθήκε τη ΔΟΕ. Μαζί με λοιπόν τι σχετικέ ε, και με την ΕΤΟΚ θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι το Βιετνάμ θα θερήσει τις δεσμεύσεις του για τις εγχώριες, τις εθνικέ ομάδες, ε, τις ομάδες. Θα έχουμε μία δική μας ομάδα η οποία θα μεταβεί στο Βιετνάμ την άλλη εβδομάδα για να προετοιμάσει το Βιετνάμ σε ό,τι αφορά το θέμα των εγχώριων αυτών ομάδων, συμβουλευτικών ομάδων, πολύ πριν από την ημερομηνία εφαρμογή, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να διδάξουμε με τι εμπειρίε μα στο Βιετνάμ. Η Πρόεδρο Φοντερ Λάιεν ανακοίνωσε επίση ότι θα υπάρξει ένα σχετικό αξιωματούχο, ο οποίο επίση θα εξετάσει πολύ ενδελεχώ τα θέματα τη υλοποίηση ε, τη Συμφωνία Ελευθερίου Εμπορίου με τον Βιετνάμ. Σε ό,τι αφορά το εμπορικό ε, έλλειμμα, ακούστηκαν κάποιοι αριθμοί και ε, προκύπτει λοιπόν αυτό το εμπορικό έλλειμμα από τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι με την θέση της εφαρμογή του της FTA θα υπάρξει μεγάλες εισαγωγές από το Βιετνάμ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, αγνόησης του κανόνων, των κανόνων της ε, προέλευσης, είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Βιετνάμ σε ό,τι αφορά την παράκαμψη αυτή των κανόνων, ε, σε ό,τι αφορά το χάλιβα, το αλουμίνιο από το Βιετνάμ. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μας δίνει ωστόσο τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και σε ό,τι αφορά το πρωτοκόλλο αμοιβαίας διοικητικής αρρωγής, όπου μπορούμε να ορίσουμε την προέλευση των προϊόντων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόσουμε και να επιβάλλουμε κυρώσεις, αν είναι αυτό απαραίτητο, για την προστασία των δεδομένων. Είναι μια συμφωνία όχι πολύ πολύ παλιά, αλλά όχι και πολύ καινούργια σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων στις FTAs. Αλλά ο αρμόδιος υπουργό από πλευρά του Βιετνάμ προγραμματίζει να νομοθετήσει στην κατεύθυνση αυτή και της σε την τεχνογνωσία μας. Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία παρέχει λοιπόν υποστηρίξη μέσω σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων σε ό,τι αφορά τον τομέα τη προστασία των δεδομένων για να μπορέσει το Βιετνάμ να νομοθετήσει προ την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά τους πόρους για την ανάπτυξη δυναμικού. Θα ξέρετε το προγράμματα που έχουμε, Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν τέτοια προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν, έχουμε και προγράμματα για τα FTI, έχουμε και διάφορες δραστηριότητε τις οποίες υποστηρίζουμε στην ΔΟΕ και πολλές ε, ΜΚΟ οι οποίε θα μας βοηθήσουν σε ό,τι αφορά την υλοποίηση ε, της συμφωνία Ελευθερίου Εμπορίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος και θέλετε να συνοψίσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα καθυστέρησε και πτήση μου από την Πράγα στι Βρυξέλλε. και αυτό ήταν ε, πέραν από τις δυνάμεις μου. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για την σημερινή τους σύμβολη και πραγματικά ελπίζω να ήταν να άξιζε τον κόπο αυτή η δελαγή απόψε. Να ακούσαμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το πώ έχει η πραγματικότητα σήμερα στο Βιετνάμ. Είμαστε προφανώ στο επίκεντρο τη προσοχή ε, σήμερα και οι δύο συμφωνίε προσεγγίζουν την τελική του φάση. Μετά την ε, κοινοβουλευτική λοιπόν έγκριση θα είναι η πρώτες τέτοιες συμφωνίες εμπορικές τόσο μεγάλης εμβέλειας στην ε, θετία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ω προ τον αντίκτυπο, είναι τεράστιε αυτές οι συμφωνίε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο, λοιπόν, τον οικονομικό, τον γεωπολιτικό, τον κοινωνικό. Ίσως να μην είμαι αμερόληπτος, γιατί το δικό μου καθήκον ως εισηγητή είναι εύκολο να κλείσουμε λοιπόν τη συμφωνία αυτή και να εξασφαλίσουμε να εγκριθεί και να υπάρξει σωστή πλειοψηφία υπέρ της συμφωνίας. Θα κάνω ό,τι μπορώ λοιπόν, ό,τι περνάει από το χέρι μου. Εκφράσατε κάποια από εσά ανησυχίε για κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την νομοθετική την εργασία και νομοθεσία, τη θέση των συνδικάτων, τον κοινωνικό διάλογο. Ακούσαμε πολλά από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την μακρά ιστορία διάδρασης με το Βιετνάμ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό μας έδωσε κάποιες καινούργιες απτικές υπό τις οποίες μπορούμε να εξετάσουμε την κατάσταση. Έγινε μια συνάντηση την τελευταία εβδομάδα μας και όδησες για να καταρτιστεί α, Ζητήθηκε να καταρτιστεί μια επιστολή προ τι Βιετνέ μαζικέ αρχέ και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα οδικό χάρτη, ένα roadmap. Θα το κάνουμε λοιπόν αυτό προφανώ αλλά από την άλλη να έχουμε υπόψη μας ε, ότι πρόκειται κυρίως για μια συμφωνία συνθήκη εμπορική, επενδυτική. Δεν ε, είναι ένα εργαλείο για να ανατραπεί το πολιτικό καθεστώς ε, στο Βιετνάμ. Μπορεί κάτι να αλλάξει και είμαστε φυσικά, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι διαφορετικό το πολιτικό σύστημα στο Βιετνάμ. Εγώ και οι συνάδελφοί μου ζούσαμε σε ένα παρόμοιο σύστημα πριν από κάποιο καιρό δεν έχει περάσει και τόσο πολύ καιρό. Καταλαβαίνω λοιπόν και κατανοώ τι ε, εσωτερικέ δυναμικέ και τι ε, ιδιαιτερότητε του συστήματο. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιου είδου συμφωνίε θα πρέπει να προωθούνται από πλευρά μα. Και πιστεύω ειλικρινά ότι οι συμφωνίε ελευθερίου εμπορίου θα βελτιώσουν τι βιωτικέ ε, συνθήκε του κόσμου του Βιετνάμ, θα δώσουν πιο πολλέ ελευθερίε και θα επιφέρουν μεγαλύτερη εμπορική ισορροπία και θα δώσουν επίση και ε, ευκαιρίε επενδύσεων στις ευρωπαϊκές εταιρείε. λαμβάνοντα υπόψη όλε τι διεθνεί δεσμεύσει του Βιετνάμ, οι οποίε προφανώ και θα πρέπει να τηρούνται. Κλείνοντα λοιπόν να πω ότι το Βιετνάμ πιστεύω ότι αλλάζει προ το καλύτερο. Έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία τις τελευταίες δεκαετίες, να το αναγνωρίσουμε αυτό, να το ενθαρρύνουμε, να ενθαρρύνουμε τη χώρα να συνεχίσει στο δρόμο αυτό και να εγκρίνουμε και τις δύο αυτές συμφωνίες, την FTA και την API, θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τα εκφράσουμε όλα αυτά. Ελπίζω λοιπόν να κάνουμε και άλλες τέτοιες συζητήσεις. Θα συνεχίσουμε αύριο, θα γίνει και μια συζήτηση μεταξύ σκιωδών και αν δεν κάνω λάθος και το Δεκέμβριο στην ε, Ολομέλεια του Στρασβούργου. Ας ε, δουλέψουμε λοιπόν σκληρά για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σίγουρα ένα μεγάλο βήμα είναι και η υιοθέτηση του εργατικού κώδικα που συζητήσαμε εδώ και φυσικά το θέμα της εφαρμογής και θα το παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγης. Εκ νέου, ευχαριστώ πολύ το επιμελητήριο. Ε, πραγματικά ήταν πολύ άριθμη αντιπροσωπή από το ΑΝΟΗ και από το Χοτσιμίνγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη ΔΟΕ. Και εσείς ήρθατε από το Βιετνάμ και καλή τύχη για τις συζητήσεις σας με την κυβέρνηση για τη διαδικασία της εφαρμογής. Και ευχαριστώ πολύ και την ITUC, την Διεθνής Ομοσπονδία Συνδικάτων. Αύριο το πρωί θα έχουμε τη συζήτηση της έκθεσης του εισηγητή και συνεχίζουμε τη διαδικασία αυτή με την Συμφωνία Εμπορίου. Σας ευχαριστώ και ολοκληρώνουμε εδώ το σημείο 6. Okay. Our next item is the item 7. And I hope that we can discuss item 7 in a Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7 σε μια ήσυχη ατμόσφαιρα, σε ένα ήσυχο κλίμα για να μπορέσουν όλοι να μιλήσουν και να Και να ακούσουν. Και αν θέλετε να συζητήσετε περιθέρετε για το θέμα του Βιετνάμ, παρακαλώ, εκτός εθούσης. Α, The ε, Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Αφορά την εφαρμογή του κανονισμού κατά των βασανιστήριων. Μία από τις επιτυχίες της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας όπου πραγματικά τονίσαμε το θέμα της εμπορικής μας πολιτικής ε, και απαγορεύσαμε την εξαγωγή κάποιων αγαθών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια. Από το 2016 εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός και θα αναθεωρηθεί το 2020 Επομένως, ε, πρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητα του κανονισμού αυτού. Έχουμε μαζί μας τη Χίλτα Χάτερμαν, που είναι επικεφαλής ε, της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για το μέσο εξωτερικής πολιτικής που θα μας μιλήσει σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού. Θα σας δώσω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που μπορώ να σα παρουσιάσω τον κανονισμό μα κατά των βασανιστήριων. Θα ήθελα να σα αναφέρω τι είναι και ποια αποτελέσματα έχει και πώ θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα και να αναφερθώ και στον κανονισμό σε παγκόσμιο πλαίσιο. Αυτός ο κανονισμό, όπω είπατε, υιοθετήθηκε το 2005 και τέθηκε έθεσε σε εφαρμογή τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλείψει τα βασανιστήρια και τη θανατική ποινή και να προωθήσει αυτό το στόχο παγκοσμίω. Ε, η κοινότητα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, έχει επενέσει το σύστημα τη Ένωση και το έχει συστήσει ω μοντέλο για τι άλλε χώρε. Ο κανονισμό αυτό κάνει δύο πράγματα. Καταρχήν, απαγορεύει την εξαγωγή ή την εισαγωγή της στην Ένωση, τη διαμετακόμιση ε, αντικειμένων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικά παρά για τη θανατική ποινή ή τα βασανιστήρια και δεύτερον για αγαθά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, για ερευνητικούς σκοπούς αλλά μπορεί να έχουν και άλλες νόμιμες χρήσης, ο κανονισμός ε, απαιτεί πρώτερη άδεια εξαγωγής. Επίσης, ο κανονισμός ε, παραθέτει προορισμούς όπου ε, πρέπει να υπάρχει γενική άδεια εξαγωγής, γιατί αυτές οι χώρες ή περιοχές έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα και έχουν αναλάβει διεθνή δέσμευση για την κατάργηση. Φυσικά, ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις αρμόδιες αρχές στα κρατη και από την τελευταία τροποποίησή του 2016, ο κανονισμός επίσης συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες για τον έλεγχο των εξαγωγών για ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε, σε ενέσεις, θανάσιμες ενέσεις στις ΗΠΑ και επίσης έχει εισαγάγει και την συντονιστική ομάδα κατά των βασινιστήριων όπου αντελάσσονται απόψεις μεταξύ κρατών μελών εμπειρογνωμόνων και επιτροπής. Τώρα, πώς αυτός ο κανονισμός παρουσιάζει αποτελέσματα και προς τα που οδεύουμε. Δύο πρόσφατες εκθέσεις που δημοσίευσε η Κομισιόν μας δείχνουν ότι αυτός ο κανονισμός γενικά εφαρμόζεται ορθά από τα κράτη-μέλη. Και ε, είναι ε, πάρα πολύ σημαντική η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών της φαρμακοβιομηχανίας και των ΜΚΟ, όπως η Διεθνής Αμνηστία, ε, η Omega Research ε, και άλλοι. Τώρα, πού πάμε από εδώ και πέρα. Φυσικά, δεν ε, μπορούμε να φυσικαζόμαστε. Και γι' αυτό σήμερα κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής και των πρακτικών ως μέρος μιας συνεχιζόμενης αναθεωρήσης του κανονισμού. Ιδίω θα εξετάσουμε τις απαιτήσει για την υποβολή εκθέσεων της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές στα κρατη και την ανάγκη για πιθανή καθοδήγηση σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες πτυχές για την εφαρμογή. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας αναθεώρησης, η Κομισιόν ε, θέλει να έχει έναν επικοδομητικό διάλογο, κυρίως μαζί σας, με το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Τέλος. Πριν να κλείσω, να πω δύο λόγια για τις σχετικές εξελίξει παγκοσμίω. Ο κανονισμός κατά των τη ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο σημαντικό καθεστώ ελέγχου που εφαρμόζεται ευρέως για αυτά τα ε, αγαθά. Όμω, πέρα από το πόσο αποτελεσματικό είναι ο οικονομισμό τη Ένωση, είναι σαφέ ότι μόνο ένα διεθνέ μέσο θα μπορούσε να καλύψει το κενό και να θέσει τέλο στο εμπόριο αυτών των φρικτών αντικειμένων. Γι' αυτό το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αργεντινή τη και τη Μογγολία ξεκίνησε την Παγκόσμια Συμμαχία ε, για το εμπόριο απελευθερωμένο από τα βασανιστήρια και τον ε, Ιούνιο του 2019 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε σημαντικό ψήφισμα που προετοιμάζει μελλοντική εργασία σε επίπεδο ΟΗΕ προς το να θεσπιστούν κοινά διεθνή πρότυπα στον τομέα καλεί το ψήφισμα να εξετάσουμε ε, το ύψε παραμέτρους, στο πεδίο εφαρμογή ε, και το εφικτό του να υπάρχουν διεθνή πρότυπα για το εμπόριο σχετικών αντικειμένων. Η Κομισιόν χρηματοδοτεί ε, το έργο της είπα της εκπροσώπου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης διερευνά το θέμα της κοπιμότητας μιας πρωτοβουλίας στον τομέα αυτό. Εμείς από την πλευρά μας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε την εισαγωγή και την ενδυνάμωση πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόμοιων εμπορικών μέτρων όπως η δική μας νομοθεσία κατά των βασανιστήριων και θα δράξουμε την ευκαιρία τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση για να διασφαλίσουμε ότι η δική μα νομοθεσία παραγμένει αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση των ασθενιστήριων και τη θανατική ποινή. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ερωτήσει. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να αναδείξω τη σημασία αυτού του κανονισμού. Πρόκειται για ένα κανονισμό που πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε. Μας κόστισε πολύ να πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις ε, προκειμένου να τεθεί σε αποτελεσματικότητα και θεωρώ ότι αποτελεί ένα νομοθετικό μέσο ε, που αποτελεί σημείο αναφορά σε διεθνές επίπεδο σήμερα. Όμως, ε, Τώρα, η έκθεση που μας παρουσιάζει το πώς ανταποκρίθηκαν τα διάφορα κράτη-μέλη μας ε, λέει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος που δεν μας έδωσε καμία πληροφορία σε σχέση με το πώς ε, λειτουργεί ο κανονισμός. Θα ήθελα να μου πείτε Ποια μέτρα έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αποφύγει να συνεχίζεται ε, μια τέτοια κατάσταση και προκειμένου όλα τα κράτη-μέλη να παρέχουν τις πληροφορίες τις οποίες έχουν δεσμευτεί να παρέχουν βάσει του κανονισμού. Επίση, θεωρώ θεμελιώδη την Παγκόσμια Συμμεχία για το εμπόριο που είναι απελευθερωμένο από τα βασανιστήρια. Γιατί καθώς αποτελεί παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αν δεν υπάρχει ε, ένας διεθνής κανονισμό, αυτό ε, μας διευκολύνει για να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε το εμπόριο τέτοιων αντικειμένων. Και πραγματικά χαίρομαι που ε, έχουμε τον αριθμό των 60 χωρών και κάθε φορά αυξάνεται ο αριθμός αυτό, αυτός. Όμως, με ανησυχεί το γεγονό ότι η επιστολή που έστειλε η κυρία Φοντελέν στον Επίτροπο Χόγκαν, όπως και στην ίδια την ακρόαση του κυρίου Χόγκαν, δεν έγινε καμία αναφορά σχετική. Ποια θα είναι η δέσμευση της Κομισιόν για να συνεχίσει να εργάζεται έτσι ώστε ο συνασπισμός αυτός ε, να ε, μπορέσει να εναγκαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χωρών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρουσίαση και σαν ομάδα είμαστε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης αυτών των προϊόντων βασανιστήριων. Αλλά το ίδιο και ε, υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της οποιασδήποτε διαφήμισης αλλά και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχω μία πιο συγκεκριμένη ερώτηση να σας κάνω. Στην έκθεση, στο 3.3 σημείο, διαβάζω το θέμα της επιβολής και κάπου λέτε ότι ίσως να μην διαθέτουμε αρκετά μέσα για την πλήρη εφαρμογή αυτών ε, των μέτρων. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να μου δώσετε τη δική σας ε, αξιολόγηση όσον αφορά τις επιπτώσεις των αποφάσεων κάποιων ε, επιχειρήσεων για την επανεγκατάσταση του κάπου αλλού, είτε σταμάτησε εντελώς η παραγωγή αυτών των προϊόντων. Κυρία Χάρντεμαν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Να απαντήσω πρώτα στην ερώτηση που αφορά τη μία χώρα. Ναι, υπάρχει μία χώρα, η Γερμανία, η οποία δημοσιεύει μια έκθεση που εξηγεί ακριβώς πώς υλοποιεί την, τον κανονισμό. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία σε αυτό που ζητάμε, αλλά βεβαίως μια επίσημη δημοσίευση, δημοσίευση μιας έκθεσης είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό από την άποψή μας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ένας τρόπος να δίνονται τα στοιχεία δημόσια. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πολύ ακριβή και συγκρίσιμα στοιχεία από μέρους των κρατών μιλών. Τώρα, τι γίνεται όσον αφορά την ολοκληρωμένη δράση και αν μπορούμε να υιοθετήσουμε διεθνή πρότυπα. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι μια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως υπάρχει αυτή η διεθνή συμμαχία. Εμείς δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε τέτοια στήριξη, ιδιαίτερα από τη Γενική Συνέλευση των ε, Ηνωμένων Εθνών. Μας στηρίζουν σήμερα πολλές χώρες, πολύ περισσότερες από αυτό που περιμέναμε. Συνεχίζουμε βεβαίως από μέρους της Προέδρου της Επιτροπής προς τον Επίτροπο Χόγκαν αλλά και όσον αφορά τη δράση που θα μπορούσε να έχει ο εκπρόσωπος ε, της εξωτερικής δράσης, ο κύριος Μπορέλ, αλλά και αυτά που μέχρι τώρα έχει κάνει η κυρία Μογκερίνη. Περιμένουμε περισσότερη δέσμευση. Δεν έχω ακόμα αν θέλετε, συζητήσει το θέμα αυτό με τον κύριο Μπορέλ, ο οποίο είναι και ο ε, άνθρωπος τον οποίο εγώ θα πρέπει να αναφερθώ για τη μέχρι τώρα δράση μας. Τώρα, όσον αφορά την απαγόρευση της ε, οποιασδήποτε διαφήμισης ε, που αφορά αυτά τα προϊόντα, βεβαίως αυτό και είναι κάτι που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, υπάρχουν όμως πάρα πολλοί περιορισμοί. Ο κανονισμός ε, αυτός βεβαίως ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ισχύει για τις εμπορικές συναλλαγές, ισχύει και για τις ε, συναλλαγές στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η πρώτη κατηγορία προϊόντων, δηλαδή προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, και για άλλους σκοπούς πέραν της ε, θανατικής ε, ποινής και των βασανιστήριων. Είχαμε επαφή με τις γαλλικές αρχές διότι η κατάσταση, αν θέλετε, όσον αφορά τη γαλλική νομοθεσία δεν ήταν σαφής. Ήρθαμε λοιπόν σε άμεση επαφή με τις γαλλικές αρχές για να διαλευκανθεί η υπόσταση και να αναλάβουν δράση οι γαλλικές αρχές. Το θέμα τώρα της διαφήμισης που αφορά τη δεύτερη κατηγορία προϊόντων. Αυτές οι κατηγορίες ε, ουσιαστικά αφορούν προϊόντα και αγαθά που έχουν και κάποια άλλη δράση, όπως παραδείγματος χάνει ιατρική χρήση. Πρόκειται για, αν θέλετε, μία ενημέρωση η οποία θα πρέπει να στοχεύει φορείς που αφορά αυτή η συγκεκριμένη χρήση, η ιατρική χρήση παραδείγματος χάνει. Κάνατε μια ερώτηση που, κύριε Πρόεδρε, που αφορά την ε, μεταφορά κάποιων επιχειρήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για να αποφύγουν τις επιπτώσεις ε, του κανονισμού αυτού. Εμείς πραγματικά συμμετέχουμε με όλες τις χώρες αυτές τις οποίες ενδεχομένως μπορεί να εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις που παράγουν αυτά τα προϊόντα. Υπάρχουν όμως και άλλοι φορείς, πέραν δηλαδή των εθνικών αρχών των χωρών αυτών, που ελέγχουν την δράση αυτών των επιχειρήσεων και αν παράγουν <clears throat> προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για νόμιμη χρήση. Ιδιαίτερα για την πρώτη κατηγορία ε, αγαθών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για φασανιστήρια ή θανατική ποινή. Υπάρχει λοιπόν εδώ η απέτηση από μέρους ε, των ε, ευρωπαϊκών αρχών να μην εξάγονται, να μην εισάγονται και να μην περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλήρης απαγόρευση λοιπόν. Και εξετάζουμε μάλιστα και την ε, πιθανότητα να απαγορευθεί η οποιαδήποτε τεχνική στήριξη αλλά και το μάρκετινγκ, η ενημέρωση και η διαφήμιση και σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης και θα χρειαστεί να περιμένουμε 10 λεπτά για να ξεκινήσουμε μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών.